E, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ε, σημερινή σύνοδο, κυρίσω την έναρξη. Θέλω να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο Φων Ρόμποϊ, να καλωσορίσω επίσης τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον επίτροπο που είναι μαζί μας. Και να περάσουμε στο πρώτο σημείο τη μερική διάταξη για σήμερα που είναι τα συμπεράσματα από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Φον Ρόμπο. Κύριε Πρόεδρε. Mr. President, uh, President of the European... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι βουλευτές. Μέσα σε 49 ημέρες προέδρευσα τριών συνεδριάσεων καθώς και τη συνεδρίαση ε, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οικονομικό και σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και επίγουσες επίσης δείχνει ότι οι συναντήσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν αποτελούν απλά μια εκδήλωση, αλλά είναι τμήμα μιας διαδικασίας. Πράγματι, στην συνεδρίαση για την οποία θα σας αναφέρω σήμερα, δηλαδή τη συνεδρίαση τη 24 η και 25 η Μαρτίου, εγκρίναμε ένα πολύ σημαντικό πακέτο μέτρων τα οποία είχαν προπαρασκευαστεί και συζητηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Αναβαθμίσαμε τη δράση μας σε σχέση με τα γεγονότα στη Λιβύη και ξεκινήσαμε, δρομολογήσαμε την απάντησή μας στις ε, καταστροφικές ε, ε, στα καταστροφικά γεγονότα της Ιαπωνίας. Θα τα αναφέρω ένα-ένα αυτά τα θέματα. Πρώτα απ' όλα, οικονομικά μέτρα. Για τα οικονομικά ζητήματα όπως είπα προωθήσαμε μια μια θέση μέτρων. Και στην ε, Σύνοδο Κορυφής ε, της Ευρωζώνης στις 11 Μαρτίου αλλά και σε άλλες συναντήσεις Ολοκληρώσαμε τελικά όλη αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, για έγκριση μέτρων και διαδικασιών για την αντιμετώπιση της κρίσης, αυτό καθ' αυτό δεν ε, οδηγεί σε έξοδο από την κρίση αυτομάτως, αλλά απαιτεί επιμονή, απαιτεί συνεχείς προσπάθειες. Δεν θέλω να επαναλαμβώ όλες τις αποφάσεις σε λεπτομέρειες, μπορείτε να τις βρείτε στα συμπεράσματα. Απλά εγώ θα ήθελα να συνοψίσω έξι σημαντικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, τροποποίηση τη συνθήκη ώστε να υπάρχει πλήρη ασφάλεια δικαίου για το μόνιμο μηχανισμό στήριξη. Στο κοινοβούλιο σα ήδη στο ψήφισμα τη 15η ε, Δεκεμβρίου είχε ζητήσει μια τροποποίηση συνθήκη που να παράσχει νομική βάση για το μηχανισμό. Αλλά όχι μια βαθιά τροποποίηση τη συνθήκης μια ελαφρά τροποποίηση. Και την συμβουλή αυτή του Κοινοβουλίου την ακολουθήσαμε. Και με ικανοποίησε ιδιαίτερα όταν εγκρίθηκε με τόσο μεγάλη πλειοψηφία στις 23 Μαρτίου η πρόταση αυτή για τροποποίηση της ε, συνθήκης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτύχαμε και διαβεβαιώσαμε το ε, Κοινοβούλιο ότι θα διασκεδάσουμε τι ανησυχίε που είχαν γερθεί για το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω του συζητητέ Μπροκ και Γκουαλτιέρη που συνεργάστηκαν εκ του σύνεγγυ μαζί μου για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματο. Δεύτερον, αναλυτική συμφωνία για το μέγεθο εύρος και τρόπο εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης του μόνιμου αλλά και βελτίωση του προσωρινού. Τρίτον, εγκρίναμε τη θέση του Συμβουλίου για έξι νομοθετικέ προτάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική μακροοικονομική εποπτεία ανώψη των ε, διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι και εσεί εργάζεστε σκληρά για το θέμα αυτό. Έχω συναντήσει του συζητητέ σα, θα του συναντήσω απόψε, θα συναντήσω μάλλον απόψε και του συντονιστέ. Οι ανησυχίε σα ε, ε, είναι και δικές μας. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τον Ιούνιο. Τέταρτον, έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρόκειται για μια άσκηση όπου παρακολουθούμε την υλοποίηση της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, το Σύμφωνο ε, Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στη μακροοικονομική εποπτεία. Τον Ιούνιο το Συμβούλιο θα καταλήξει στα δέοντα συμπεράσματα και εγώ προσωπικώς θα φροντίσω να μην μεταβληθεί αυτό σε μια απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Πέμπτον, θα πρέπει να γίνουν αξιόπιστες δοκιμές αντοχής για τις τράπεζες. Διπλό το καθήκον και θα πρέπει να γίνει αυτή η δοκιμή από τις τράπεζες αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει σε κάθε χώρα να αντιμετωπίσει και να ε, προβεί στα απαραίτητα μέτρα. Επίσης, συντονισμός έκτος. Ε, το πακέτο ε, ευρώ συν Φυσικά και οι χώρες Ευρωζώνης θέλουν να, αναλάβουν ακόμα μεγαλύτερες ε, δεσμεύσεις αλλά και οι υπόλοιπες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν. Έξι χώρες που δεν είναι στο ευρώ έχουν ήδη ανακοινώσει ότι σε αυτό το σύμφωνο θα, θα συμμετάσχουν ε, Δανία, Πολωνία, Λετωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία και βέβαια οποιαδήποτε άλλη από τις τέσσερις εναπομένουσες χώρες μπορεί να συμμετάσχει. Θέλω να πω ότι η πολιτική δέσμευση αυτού του πακέτου ε, ευρώ-συν είναι συμπληρωματικό ε, σε όλη την υπόλοιπη δέσμη μέτρων για ενίσχυση του πακέτου για τη χρηματοοικονομική εποπτεία, τη μακροοικονομική εποπτεία, την εφαρμογή της σημαντικής στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τη στρατηγική μεταρρύθμιση για την οικονομική ανάπτυξη. Οι δεσμεύσει σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, δημόσια οικονομικά, συντάξει, απασχόληση κτλ. θα πρέπει να μεταφραστούν ε, σε εθνικά προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης, τα οποία θα αξιολογούνται ετησίως στο ανώτατο επίπεδο. Και μια τελευταία παρατήρηση για την οικονομία. Ίσως ορισμένοι φοβούνται ότι ο στόχος είναι να υποβαθμιστεί το κοινωνικό κράτος σε καμία περίπτωση. Ο στόχος είναι ακριβώς ο αντίθετος, να εξασφαλίσουμε, να ε, διασώσουμε αυτό το μοντέλο. Θέλουμε οι οικονομίες μας να είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να μπορούν να διατηρήσουν ε, το, ε, την ευημερία όλων των πολιτών. Περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό εργαζόμαστε. Αυτά λοιπόν τα βασικά στοιχεία του πακέτου οικονομικών μέτρων για να μπορέσουμε να εξέλθουμε από την κρίση. Όπως είπα, Πρόκειται για προϊόν μακράς διαδικασίας, όχι προϊόν μίας και μόνης συνεδρίασης. Στις 25 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να βελτιώσει την οικονομική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ξεκίνησε τις εργασίες της ε, η ομάδα εργασίας της οποίας προείδευα. Και ένα χρόνο μετά είχαμε νέους κανόνες, νέα εργαλεία και πιο φιλόδοξες πολιτικές. Ήταν και παραμένει προσπάθεια όλων των θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου και όλων των κρατών μελών. Δεν είναι πάντοτε εύκολο το εγχείρημα. Κάποτε είναι συναισθηματικά φορτισμένη όλη η προσπάθεια, αλλά στόχος είναι να έχουμε μια σαφή κατεύθυνση και να επιτύχουμε αυτά αποτελέσματα. Ήδη έχουμε αποτελέσματα, φυσικά δεν έχουμε ε, ξεπεράσει όλα τα προβλήματα, διότι αυτά αποτελούν προϊόν παλαιών ε, σφαλμάτων και ελλείψεως ε, μέσων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα όμως γνωρίζουμε ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να μην επαναλάβουμε τα ασφάλματα του παρελθόντος. Έρχομαι στη Λιβύη. Φυσικά στις 24 και 25 Μαρτίου συζητήσαμε και για την κατάσταση στη Λιβύη και δείξαμε ότι είμαστε αποφασισμένοι από κοινού. Ορισμένοι από εσά ξέρω ότι έχετε αμφιβολίε. Πάντω, εργαστήκαμε σκληρά για να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πριν από δύο εβδομάδε, σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στι 11 Μαρτίου, είχαμε καθορίσει μια κοινή γραμμή. Και έπειτα αν δεν ε, υπήρχε αυτή η γραμμή δεν θα μπορούσαμε να λάβουμε τις συγκεκριμένε αποφάσεις. Είπαμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, την ασφάλεια των πολιτών της Λιβύης και θα εξετάσουμε όλες τις επιλογές, αλλά μόνο αν υπάρξει σαφής ανάγκη, αν υπάρξει σαφής νομική βάση και ανάγκη στήριξης της περιοχής. Αυτές οι προϋποθέσεις ε, συνέτρεχαν, ήταν σαφές αυτό όταν είδαμε ότι το καθεστώς κάνει όλο και μεγαλύτερες ε, επιθέσεις κατά του ίδιου του πληθυσμού της χώρας. Ε, ο Αραβικός Σύνδεσμος μας υποστήριξε ανέλαβαν δράση οι σύμμαχοι από τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τις αραβικές χώρες με στόχο να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό της Λιβύης ώστε να αποφευχθεί όπως και απεφεύθη μια ε, αιματοχυσία. Πραγματικά ε, σώθηκαν χιλιάδες ζωές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα που δείχνει την ύψιστη προσοχή που δίνουμε και βέβαια και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, διότι το δάσος είναι σημαντικότερο από το δέντρο ή τα δέντρα. Βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι η απόφαση για ανάληψη στρατιωτικής δράσης δεν ήταν εύκολη. Φυσικά υπήρχαν ερωτήσεις, υπήρχαν ε, καχυποψίες και δισταγμοί Υπάρχει αυτό το θέμα του πολέμου κίνησης, αλλά οποιαδήποτε δυσκολία που έχουμε αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της πτυχής αυτής της κρίσης δεν θα πρέπει να συγκαλύπτει σε καμία περίπτωση την, το όλο ιστορικό των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτής εξ αρχής είμαστε στην πρώτη γραμμή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα επιβάλλουμε κυρώσεις. Πρώτη, επιβάλαμε απαγόρευση ε, μετακίνηση σημαντικών προσωπικότητων, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων. Αναγνώρισαμε πρώτη επίση ω έγκυρο συνομιλητή μα ε, το Εθνικό Συμβούλιο και επίση συντονίσαμε τι προσπάθειε διάσωση ε, και απεκλωβισμού των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζουμε να παρέχουμε σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια. Οι πολιτικοί στόχοι που θεσπίσαμε στι 11 Μαρτίου δεν έχουν αλλάξει. Ο Καντάφη θα πρέπει να φύγει και εμεί θέλουμε μια πολιτική μετάβαση μετάβαση, τις οποίες θα ηγηθούν οι ίδιοι οι Λίβοι βάσει του πολιτικού διαλόγου. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε για μια νέα Λιβύη και οικονομικά αλλά και σε ό,τι αφορά ε, την οικοδόμηση των νέων θεσμών Τη Επίσης παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και τα γεγονότα στην υπόλοιπη, στην ευρύτερη περιοχή. Η κατάσταση είναι διαφορετική σε κάθε χώρα. Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση στη Συρία, την Ιεμένη και τον Μπαχρέιν. Καταδικάζουμε την κλιμάκωση της βίας και στηρίζουμε τις πολιτικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τις πολιτικές μας και θα συζητήσουμε αργότερα με αρκετά μέλη που είναι αρμόδια για την ευρύτερη αυτή περιοχή τα σχετικά στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Τώρα κάτι θετικό ομαλή διεξαγωγή ε, του συνταγματικού ε, δημοψήφισματος πριν από δύο εβδομάδες στην Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά την ακτή ελεφαντοστούν από δύο λόγια, δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη ε, του πιο πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εγκρίναμε ωστόσο συμπεράσματα το Δεκέμβριο και παρακολουθούμε και του σύνεγγυς της εξελίξης εκεί έκτοτε. Πρώτα απ' όλα καταδικάζουμε τη βία ιδιαίτερα την βία κατά αμάχων. Αυτό ε, είναι απερίφραστο. Απερίφραστη δίκη της βίας και πρέπει να σταματήσει από όλες τις πλευρές. Δεύτερον, η τρέχουσα κατάσταση είναι ένα σαφές αποτέλεσμα της έλλειψης σεβασμού στη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν αφορά τις εκλογές μόνο, ε, είναι ο σεβασμός και το αποτελέσμα των εκλογών. Η διεθνή κοινότητα ήταν σαφής για το αποτέλεσμα των περσινών προεδρικών εκλογών στην ακτή του. και θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς στην απόφασή μας. Σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία τέλος, και σε ό,τι αφορά τη συσσόρευση αυτών των τραγωδιών που έπληξαν ε, την Ιαπωνία. Εκφράζουμε ε, τη συμπάθεια, την αλληλεγγύη μας ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς το λαό της Ιαπωνίας, αλλά και τα συλληπιτήριά μας για τις χιλιάδες ε, θυμάτων. Δεν το λησμονούμε αυτό, παρότι υπάρχουν και άλλες πτυχές της Ιαπωνικής τραγωδίας που έχουν επισύρει την προσοχή μας. Όπως μπορούμε, με όποιο τρόπο μπορούμε θα βοηθήσουμε τους φίλους μας από την Ιαπωνία διότι είναι πολύ σημαντικέ οι σχέσει μεταξύ Ιαπωνία-Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι υπερβαίνει την Ιαπωνία το αποτέλεσμα αυτή τη ε, κατάσταση και εμεί ε, αντλούμε τα διδάγματα ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε τι συνέπειε θα έχει η κρίση αυτή και για την παγκόσμια οικονομία και σε ό,τι αφορά όμω ε, την ατομική, την πυρηνική ενέργεια, που είναι πολύ σημαντικό. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι η ασφάλεια όλων των πυρηνικών εργοστασίων μα θα πρέπει να αναθεωρηθεί κατεπηγόντω στο πλαίσιο δοκιμών αντοχή και ασφάλεια και θα υπάρξει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από το τέλη του χρόνου σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων. Θα αναθεωρήσουμε τους κανόνες ασφάλειας των πυρηνικών εργοστασίων και όπου χρειαστεί θα κάνουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη θέλουμε τα ύψιστα δυνατά πρότυπα για την πυρηνική ασφάλεια. Δηλαδή αν υπάρχει ε, ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων. Ε, σίγουρα λύνονται κάποια προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να περιοριστεί αυτό μόνο στην Ευρώπη. Χρειάζεται παγκόσμια ε, αναθεώρηση και εξέταση τη ασφάλεια όλων των πυρηνικών εργοστασίων ανά τον κόσμο. Έτσι ολοκληρώνω την ε, περιληπτική αναφορά μου στα ε, πεπραγμένα τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που σε μεγάλο βαθμό έχει ανοίξει το δρόμο και για τι νομοθετικέ διαδικασίε, αλλά και για τον γενικότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο που αποτελεί δικαίωμα του Κοινοβουλίου Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της πολιτικής ασφάλειας. Και τώρα προσβλέπω στις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, the Μετά θα ήθελα να ζητήσω τον κύριο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόσο, να πάρει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο πρόεδρος του Πολιτικού Συμβουλίου μας παρουσίασε όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την σύνοδο της περασμένης εβδομάδας. Επιτρέψτε μου να συμμεριστώ μαζί σας πώς ερμηνεύω αυτά που υπόθηκαν και να πω κάποια πράγματα για τα μελλοντικά βήματα. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι διαθροτικές σημαντικές αποφάσεις έχουν ληφθεί για μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη, καλύτερο οικονομικό συντονισμό επίσης. Είναι πραγματική καμπή για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη, κυρίως όμως σκεφτούμε το μονοπάτι που έχουμε διανύσει. Έχουμε ενοποιήσει την οικονομική Ένωση, την οικονομική πτυχή της Οικονομικής και Νομισματικής Ενώσεως και τώρα θα έχουμε σταθερότερες βάσεις πιστεύω. Διαθέτουμε πλέον ένα πλαίσιο για να δώσουμε καλύτερες απαντήσεις όλοι μαζί σε κρίσεις που θα μπορούσαν να εμφανιστούν. Και τελευταίο στοιχείο, για να εκτιμήσουμε και τα αποτελέσματα του Συμβουλίου, μπορούμε να πούμε ότι το πλαίσιο σέβεται τις διατάξεις της συνθήκης και ακολουθεί μια προσέγγιση κοινοτική. Ξέρουμε ότι αυτά δεν τα ήταν δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν στην πρώτη θέση για να δώσει απάντηση στην κρίση και για να προωθήσει την Ευρώπη στον ορίζοντα 2020. Λοιπόν, το Κοινοβούλιο μας υποστήριξε και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί μας στηρίξατε τις προσπάθειές μας. Λάβαμε αποφάσεις από κοινού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για την προάσπιση της κοινωτικής προσεγγίσεως. Εισακούστηκαν οι προσπάθειές μας και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Η νέα μας οικονομική δομή ε, έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο ποσοστό, αλλά δεν αποτελεί εχέγγυο αυτό καθε αυτό. Θα πρέπει οι πολιτικοί υπεύθυνοι να λάβουν τις ουσιαστικές αποφάσεις που απαιτούνται. Θα πρέπει στο νέο πλαίσιο με αποφασιστικότητα και χωρίς καθυστέρηση να εφαρμόσουμε τις προτεραιότητες για τις διαθεωτικές μεταρρυθμίσεις και την οικονομική εξυγίανση που απαιτούνται για την ανάπτυξη. Αποφάσεις περίπτωσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί τη βάση τη αιτήσια εξετάσεω τη ανάπτυξη ε, τη έρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω την πεποίθηση ότι η αποφασιστικότητά μα θα είναι εξίσου σημαντική στου επόμενου μήνε και τα χρόνια, όπω η αποφασιστικότητα που δείξαμε μέχρι τώρα, για να εφαρμόσουμε συντονισμένο τρόπο τα διάφορα στοιχεία ε, τη σφαιρική απαντήσεώ μα για την κρίση. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, ε, και το σύμφωνο Ευρώπλας, το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης των ισχυμένων καθώς και τα αλληλέγγυα μέτρα ε, θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη χρηματοστητική σταθερότητα της Ευρωζώνης. Δεν σας αποκρυπτώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να προχωρήσει πιο πέρα ακόμα σε αρκετούς τομείς στην οικονομική διακυβέρνηση και κυρίως ε, όσον αφορά το νέο μηχανισμό ε, οικονομικής στήριξης της Ευρωζώνης. Θέλαμε να έχουμε περισσότερη ευελιξία επί παραδείγματι. Όμως ε, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι καταφέραμε να πετύχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος εδράζεται επί της συνθήκης με ισχυρή παρέμβαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το επιτευχθένα αποτέλεσμα είναι σημαντικό και η θετική τοποθέτηση αφορά την τροποποίηση της συνθήκης που ενεκρίθη με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, βουλευτές, θα πρέπει τώρα πλέον να δημιουργήσουμε νέε δομές διακυβέρνηση προς εξυπηρέτηση απαντήσεω σε συγκυρία. Στην πραγματικότητα η συγκυρία παραμένει δύσκολη. Και τώρα το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των 100 μελών που θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα εθνικά τους μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από κάθε κάτος μέλος προτάσεις συγκεκριμένε και φιλόδοξες, ούτω ώστε να προχωρήσουμε από κοινού στο δρόμο των μεγάλων στόχων της στρατηγικής της Ευρώπης το 2020. Ήτι περισσότερη απασχόληση, περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία, στην κατάρτιση, στην έρευνα και στην καινοτομία, επίσης για την καταπολέμηση με πιο γενναίο τρόπο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Περιμένουμε επίσης και την παρουσίαση μέτρων για διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που διαρκούν και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη για την απασχόληση. Από τη στιγμή που θα λάβουμε τα έγγραφα, θα μπορέσουμε τότε να προετοιμάσουμε μια πρόταση γνωμοδοτήσεω και συστάσει κατά χώρα. Ούτω ώστε να υιοθετηθούν πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του μηνό Ιουνίου, που θα σημειώσει το τέλο του κύκλου του πρώτου εξαμήνου του Ευρωπαϊκού που θεσπίσαμε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι συμμεριζόμεθα όλοι εδώ κοινή ευθύνη και ότι είναι σημαντικό καθένας ε, να ενστερνιστεί την ε, Στατηγική Ευρώπη 2020. Αυτή η στρατηγική είναι το βασικό πλαίσιο για τις μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Και θα ήθελα εδώ ε, να αναφερθώ στο σημείο 6 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που επιμένουν και λένε και παραθέτω ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτών των πολιτικών και για να επιτευχθεί μεγάλη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία μια συνεργασία άμεση θα εξασφαλίζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά κά όργανα και όργανα συμβουλευτικά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών. Τα Εθνικά Κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι περιφέρειες και άλλοι φορείς θα εμπλακούν άμεσα. Τέλος παράθεσης. Επιμένω από αυτού, διότι ακούγονται πολύ συχνά επικρίσεις της αντικείτησης Αβώνας. Ακούστηκαν η έλλειψη του ownership ε, για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να αντλήσουμε ε, τα μαθήματα από την πρώτερη διαδικασία και αυτή τη φορά πραγματικά να κινηθούμε στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και να καταβάλουμε μια προσπάθεια σοβαρή για την ανάπτυξη, για την απασχόληση. Τώρα, όσον αφορά το μέτωπο τη μεταρρύθμιση τη οικονομική διακυβερνήσεω, τώρα εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να προχωρήσει προ την τελική έγκριση του πακέτου των έξι νομοθετικών προτάσεων και ελπίζω ότι σύντομα θα καταλήξουμε στην επίτευξη του φιλοδόξου αποτελέσματος. Είναι ουσιαστικό για να έχουμε όλο το σύστημα αυτό διακυβέρνηση που θα λειτουργεί. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλοί λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά επίσης και πολλούς λόγους για να μην φυστούμε προσπαθειών. Αντιθέτως, διότι η συγκυρία παραμένει δύσκολη και αβέβαιη, να προχωρήσουμε κυρίως όσον αφορά τι κοινωνικές πτυχές που μας ανησυχούν όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, τι επόμενε εβδομάδε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει επίση τι προτάσει τη επί τη πράξη για την ενιαία αγορά. Και θα ήθελα να πω ότι ικανοποιούμε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφιέρωσε πολύ χρόνο συζητήσει για το μέλλον τη ενιαία αγορά και ότι υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο τη ενιαία αγορά που θα τονώσει έτσι την ανάπτυξη και την απασχόληση και θα ευνοήσει την ανταγωνιστικότητα υπογραμμίζοντας τη σημασία τη μειώσεω των ρυθμιστικών περιορισμών που βαρύνουν όλους ιδιαίτερως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε λοιπόν να απελευθερώσουμε το δυναμικό τη αναπτύξεω ενία αγορά. Και θα ήθελα να επενθυμίσω εδώ ότι η διαβούλευση για τα δημοσιονομικά δεν αποτελεί έναν αυτό σκοπό, αλλά ένα μέσο για να ενεργοποιήσουμε μια ισότιμη βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση. Και όσο, εφόσον μιλάμε για ισότιμη αυτή ανάπτυξη, θα πρέπει να υπογραμμίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίση, τοποθετήθηκε επί τι δυνατότητε να υπάρχει ένα φόρο επί των συναλλαγών Φόρο επί των χρηματοδοτικών συναλλαγών των διεθνών. Και επιβεβαίωσα την πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχετικέ προτάσει στον τομέα της ως του τομέα του χρηματοδοτικού. Πιστεύουμε μάλιστα ότι θα πρέπει να ε, συμβάλλουμε και εμεί σε μια απάντηση μέσω αυτού ε, στην κρίση. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε, όπω γνωρίζετε, και την κατάσταση στη Νότια Μεσόγειο και στη Λιβύη. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρουσίασε μια έκθεση λεπτομερέστατη θα μπορούσα απλούστατα να σας αναφέρω τις συνομιλίες που είχα χτε με τον Πρωθυπουργό της Τινησίας. Επανέλαβα εγώ την υποστήριξή μας στη Δημοκρατική Επανάσταση και τη διαθεσιμότητά μας να βοηθήσουμε τον Τινησιακό λαό στην προσπάθεια που καταβάλει για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ισοτιμία και τόνισα και τα θέματα τη μετανάστευση. Ότι εκεί η Τινησία και η Ευρώπη θα πρέπει να το συζητήσουν το θέμα τη μετανάστευση από κοινού Ένα πνεύμα πραγματική εταιρική σχέσεω. Ε, σύμπραξη για τη δημοκρατία για την ευμάρεια, την κοινή ευμάρεια. Τέτοια προτείναμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, συμφώνησε με αυτά. Άλλο θέμα που απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η κρίση στην Ιαπωνία, κυρίως οι πυρηνικές πτυχές αυτής. Χθες συζήτησα τηλεφωνικά με τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό. Πάμε σημαντικά πράγματα. Εκείνος ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δράσεις της και του εξέφρασα εκ νέου την αλληλεγγύη μα και του επιβεβαίωσα ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό του. Συζητήσαμε επίση και το θέμα το πυρηνικό. Ο Πρωθυπουργό Καν με ενημερώσε για την κατάσταση που κρατεί στην Ιαπωνία όσον αφορά τι πρόσφατε εξελίξει όσον αφορά την ασφάλεια και υπογράμμισε τη διαθεσιμότητά του για τη συνεργασία μαζί μα, τι προσπάθειε που θα καταβληθούν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τα θέματα τη πυρηνική ασφαλεία. Είναι προφανέ ότι υπάρχει ανησυχία που αυξάνεται όσον αφορά τα πυρηνικά. Θα πρέπει να δοθεί απάντηση στι ανησυχίε αυτέ και να εξασφαλιστεί μια ασφάλεια μέγιστη στα πυρηνικά. Θα πρέπει να δράσουμε με πλήρη διαφάνεια. Άρα θα γίνουν δοκιμέ αντοχή των πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιφόρτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Φορέων στον τομέα τη ασφάλεια των πυρηνικών να καθορίσουν τι τάσει και λεπτομέρειε των δοκιμών που θα κάνουν οι εθνικέ αρχέ οι ανεξάρτητε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει επίση και το πλαίσιο το νομοθετικό και ρυθμιστικό που υπάρχει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των πυρηνικών και θα προτείνει μέχρι το τέλο του έτου όλε τι βελτιώσει που ίσω θα ε, πρέπει να θεωρηθούν απαραίτητε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, δεν θα πρέπει να απογοητεύσουμε τις ελπίδες που υπάρχουν για κοινή ε, προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθημερινά άοκνα εργάζεται, γνωρίζοντα ότι μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου σα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, επομιζόμενοι πλήρω τις νέε ευθύνε μα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Ντόιλα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόσμο. Κόμμα. Κύριε Πρόεδρε, πρόοδευσαν οι χώρες μας προς σωστή μετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυξήθηκε ε, η πρικοδότηση του μηχανισμού στήριξης, γίνεται μόνιμος. Δείχνουμε έτσι την αφοσίωσή μας στο ευρώ αλλά και την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών αφενός αυτών που είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και αφετέρου αυτών που αντιμετωπίζουν προσωρινά κάποιες δυσκολίες. Επίσης, ό,τι αφορά τις αποφάσεις ε, για την Ευρωζώνη, αυτό το πακέτο ΣΥΝ δείχνει επίσης ε, πόσο ε, μεγάλη είναι η πρόθεση των ηγετών της Ευρώπης να διδαχθούν από την κρίση θέλουμε να είμαστε πιο συνεπείς στις κοινωνικο-οικονομικές μας επιλογές. Έχει περάσει ο καιρός που κάθε χώρα μπορούσε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους εταίρους της ε, να ε, προβλέπει ένα άτυπο ε, φορολογικό συντελεστή ή κάποια άλλα μέτρα ιδιαίτερα για τον πολύ απλό λόγο ότι όλες οι χώρες πρέπει να χαίρουν της αλληλεγγύη των εταίρων τους. Αλλά αυτή η αλληλεγγύη θα γίνει αποδεκτή από τους λαούς μας μόνο αν γνωρίζουν ότι κάνουμε όλοι συγκρίσιμε προσπάθειες για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και του δημόσιου χρέου. Και αυτό το πακέτο είναι πολύ σημαντικό για να υπάρξει σύγκληση των οικονομιών μα. Η ομάδα μα υποστηρίζει στεναρά αυτό το πακέτο και πάντοτε όμω θα ζητούμε η εφαρμογή του να γίνει στο πλαίσιο τη κοινοτική μεθόδου υπό την αιγίδα της Κομισιόν, αγαπητέ μου Πρόεδρε. Πράγματι, επιτύχατε πρόοδο Κάνατε καλή δουλειά θα έλεγα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη με την κοινοτική μέθοδο, επαναλαμβάνω υπό την αιγέδα τη Κομισιόν. Έτσι θα οικοδομήσουμε την Ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε είμαι ε, πάρα πολύ πείσμων και ξεροκέφαλο και κάθε φορά θα το ξαναλέω αυτό, για να μην το ξεχάσετε. Λοιπόν, η Ευρώπη δεν διακρίνεται μόνο με το, με το κοινωνικό μοντέλο ε, της ε, οικονομία τη αγοράς. Είναι ένα μοντέλο στο οποίο είμαστε προσιλωμένοι και βασίζεται στην αρχή τη αλληλεγγύη. Είναι δύσκολο όμω να διατηρηθεί στο πλαίσιο τη παγκοσμιοποίηση στο μοντέλο αυτό. Επομένω, το ερώτημα που τίθεται είναι πώ θα εξασφαλίσουμε για αυτό το μοντέλο ένα βιώσιμο μέλλον, βρίσκοντα τη χρυσή τομή μεταξύ αυτού που ζητούν οι σοσιαλιστές ενό μοντέλο που μας οδηγεί στο, στην ε, χρεοκοπία αλλά και της του υπερβολικού φιλευθερισμού που επίσης μας οδηγεί ε, σε κρίση. Πρέπει λοιπόν πρώτον όλες οι χώρες να μειώσουν τα έλλειμματά τους, δεύτερον να εγκρίνουν δημοσιονομικούς, φορολογικούς, κοινωνικούς κανόνες που είναι συγκρίσιμοι και τρίτον να επενδύσουν όλες οι χώρες μαζί στην καινοτομία ώστε να έχουμε ε, περισσότερη ρακορδίλα για την ανάπτυξη, το οποίο είναι ανεπαρκή. Πρέπει να ενισχύσουμε, πρέπει να διατηρήσουμε το μοντέλο μας και αυτό θα το πετύχουμε εάν ε, επενδύσουμε στη βιοτεχνολογία, την ανοτεχνολογία, στην πράσινη ενέργεια κτλ εάν αυξήσουμε τα περιθώριά μας ή αν ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της ανάπτυξης και αν κάνουμε οικονομίες ε, κλίμακας, συγκέντρωσης ε, των κεφαλαίων και των δυνάμεών μας. Εάν δεν επενδύσουμε στην καινοτομία και αν δεν έχουμε ευρωπαϊκό όραμα, δεν θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τους άλλους ανταγωνιστές μας. Όσο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνεδρίαζαν πριν από 10 χρόνια, το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα συνέχιζε να ανισχύει ολόκληρο τον κόσμο. Και επαναστάτε ε, τη Λιβύη επίσης ζητούσαν ε, μια ισχυρή ε, ένδειξη, μια χειρονομία εκ μέρου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δείξουμε πνεύμα ευθύνη. Δείξαμε σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά πνεύμα ευθύνης δώσαμε την τεχνογνωσία μας στο πλαίσιο αυτής της πολύ ανησυχητικής κατάστασης, όχι μόνο για την Ιαπωνία αλλά και για τη διεθνή κοινότητα. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ένα πριν και ένα μετά τη Φουκουσίμα. Η ομάδα μας θα ήθελε η μετά τη Φουκουσίμα περίοδος, παρότι δεν έχει φτάσει ακόμη, να είναι μια περίοδος προβληματισμού, δράσης, αναστοχασμού, ώστε να ενισχυθούν σημαντικά οι κανόνες πυρηνικής ασφάλειας αφενός και αφετέρου να αυξηθούν οι προσπάθειές μας στον τομέα της πράσινης ενέργειας. Συμφωνώ με την προσέγγιση σας κύριε Πρόεδρε ε, σε ό,τι αφορά την ακτή του Ελεφαντοστού. Σε ό,τι αφορά τέλος τη Μεσόγειο, χαιρετίζω ε, την έκκληση που απίφθινε εκ νέου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, για απόσυρση του Καντάφη, για να, υπάρξει ένα νέα, να υπάρξουν νέα θεμέλια στη χώρα αυτή. Όλες οι χώρες θα πρέπει να υποστηρίξουν την φιλόδοξη πολιτική γειτονία, όπως αυτό έγινε για την Ανατολή τη δεκαετία του 90, να γίνει για τον Νότο σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. Μάρτιν Σούλτς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντα τι μα λένε ο κύριο ε, Φαρόμπα και ο κύριο Μπαρόσο ε, προσεκτικά, ε, μας έρχεται στο μυαλό το γερμανικό τραγούδι ότι τα έχουμε όλα υπό έλεγχο, λες και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όλα easy. Τα έχουμε λύσει όλα και έχουμε ικανοποιήσει τους πάντες. Οι παρουσιάσεις σας και η έκθεσή σας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Σας ε, κατανοώ που έρχεστε εδώ για να μην ε, και δεν μας λέτε ε, αρνητικά στοιχεία. Και εγώ αν ήμουν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν θα ερχόμουν εδώ να τα παρουσιάσω όλα αρνητικά. Αλλά μιλήσατε για τη Λιβύη. Δεν αναφέρατε όμως την βαθιά, τον βαθύ διχασμό των δύο βασικών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για το θέμα αυτό. Μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας δεν υπάρχει καμία συμφωνία σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Αυτός ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα μας καταδεικνύει ότι δεν είναι όλα υπό έλεγχο. Το αποτέλεσμα του συμβουλίου αυτού, κυρία Φαν Ρόμπαϊ, το είχαμε, θα μπορούσαμε να το έχουμε πετύχει και το 2010. Μη σας πω, θα έπρεπε να το είχαμε πετύχει το 2010, αν θέλαμε να αποτρέψουμε μια αρνητική, ένα αρνητικό φαυλοκύκλο στην Ευρωζώνη. Την άνοιξη του 2010 έπρεπε να το είχαμε κάνει αυτό. Και για θα πρέπει να ρωτηθούμε γιατί δεν το κάναμε την άνοιξη του 2010, γιατί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο θεσμικό αυτό όργανο του οποίου προεδρεύεται, δεν επικρατεί η κοινοτική μέθοδος, δεν επικρατεί το κοινοτικό πνεύμα, ο κοινοτικός στόχος, ο κοινό στόχος. Δεν καθορίζει αυτός αυτά που αποφασίζονται, όχι. Η τελευταία, αν θέλετε, εθνική αμφισβήτηση, ο τελευταίος εθνικός δισταγμός μετράει πιο πολύ από την κοινή μέθοδο. Εγώ, κυρία Μπαρόσο, θα ήθελα να είχατε μιλήσει για το πώς είναι δυνατόν το κόμμα στο οποίο ανήκετε, του οποίου ήσασταν και πρόεδρος, που σας έκανε πρωθυπουργό στην Πορτογαλία. Πώς γίνεται το κόμμα αυτό, το ίδιο κόμμα, να ρίχνει μια κυβέρνηση η οποία περνάει τα μέτρα στην Πορτογαλία τα οποία εσείς και ο διπλανός σας επίτροπος έχετε πετύσει. Αυτό δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς εσάς. Ε, ε, δεν είσαστε πλέον ε, πρόεδρος του κόμματος. Θα ήθελα όμως μία δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δεκτική αυτή κίνηση. Γιατί η πτώση της κυβέρνησης αυτής έρχεται σε μία χρονική συγκυρία όπου η κυβέρνηση αυτή επιτέλους συμφωνεί να κάνει αυτά που προβλέπουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και που απαιτεί το Σύμφωνο Σταθερότητας. Μα θα προχωρήσει έτσι η Ευρώπη, δεν είναι δυνατόν. Και αυτό που με ανησύχησε ιδιαίτερα είναι το ότι δεν άκουσα καμία κουβέντα για το εξή. Πάντα πριν από ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βλέπουμε την ίδια ταινία. Δεν συμφωνούν οι κυβερνήσεις για μέτρα σταθερότητας. Μάλλον Μόλις ε, αποφασίζουν οι κυβερνήσει για μέτρα σταθεροποίηση για μια χώρα, έρχεται ένας οίκο αξιολόγηση και υποβιβάζει τη χώρα αυτή και την αφήνει ε, θύμα στις ε, κερδοσκοπικές ε, τάσεις. Πότε θα πούμε ότι δεν θα επιτρέψουμε στην Ευρώπη να κυβερνάται από τέτοιους κερδοσκόπους. Και τι λέμε για τις τράπεζες ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ που το είπατε αυτό κύριε Μπαρόσο, ότι θα υποβάλω μία πρόταση για τον φόρο το χρηματοπιστωτικό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επί του παρόντος ε, δανείζει με 1% επιτόκιο στις ίδιες τράπεζες οι οποίες δανείζουν με 10% στα κράτη-μέλη στην Ευρωζώνη συνεχίζει η κατάσταση, γιατί αυτοί που έχουν προκαλέσει την κρίση είναι αυτοί που τελικά κερδοσκοπούν από την κρίση. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιβληθεί ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για να συμμετάσχουν στις συνέπειες Τη κρίση. Κύριε Μπαρόσο, μιλήσατε και για την Ευρώπη του 2020, για πιο πολλή απασχόληση, για επενδύσεις, πιο πολλή ε, έρευνα, ε, πιο πολλή προστασία του περιβάλλοντο. Τέλεια, αλλά όλο και πιο λίγε δημόσιε επενδύσει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι η Ευρώπη 2020 είναι φανταστικό ε, σχέδιο, όπως και η Λισαβόνα, η στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά θα αποτύχει αν συνεχίσουμε την περικόπη των προπολογισμών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι θάρρος για δημόσιες επενδύσεις. Κοιτάξτε τις επενδύσεις στις αναδυόμενες ε, χώρες. Κοιτάξτε τις δημόσιες επενδύσεις στην Ινδία, στην Βραζιλία, στις άλλες υπήρους. Τι επενδύεται από το κράτος. Η Ευρώπη ε, περικόπτει τις επενδύσεις αυτές και συμβάλλει στον ίδιο της το θάνατο και η Ευρώπη 2020 τελικά θα αποτελέσει νομική βάση και υποχρεώνεται τελικά τις κυβερνήσεις να κάνουν αυτά που εξαγγέλουν, αλλά μετά τα αποτρέπουμε όλα αυτά, μεταξύ άλλων και με την περικοπή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Γι' αυτό πιστεύω, κύριε Μπαρόσο, από εσάς περιμένω το εξής ε, και από τον κύριο Λεβαντόφσκι ένα ε, δεσμευμένο σχέδιο για ένα προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελείωσε ο χρόνος σας, διακόπτει ο Πρόεδρος. Κυρία Πρόεδρε Χι Φαρχόφστατ από τους ε, Φιλελεύθερους και Δημοκράτες. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση αυτή από πλευράς ε, του Συμβουλίου. Αλλά α είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα. Δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει η κρίση και δεν θεωρώ ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε τώρα μπορούν να βάλουν ένα τέρμα στην κρίση. α είμαστε ειλικρινεί ότι είναι μεγάλη η θύελα που επίκειται. Ω τώρα τι κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνάδελφοι, χρησιμοποιούμε μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα, δεν αντιμετωπίζουν τα αίτια της Κρήτης. Έχουμε δώσει 110 δις στην Ελλάδα. Έχουμε δώσει 67 δις στην Ιρλανδία και δεν συμπεριλαμβάνουν τα 24 δις που αποφασίσαμε να δοθούν στις Ιρλανδικές τράπεζες. Επί του παρόντος, 76 δις έχουμε δώσει κρατικά ομόλογα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει γιατί και επιπλέον έχουμε 100 δισεκατομμύρια εγγυήσει στην Ευρώπη. Μιλάμε για 400 δις αθρηστικά συνολικά. Τόσα έχουμε επενδύσει τους τελευταίους μήνες στην κρίση και αυτό είναι το τριπλάσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και δεν έχουμε δει και τα χειρότερα ακόμα. Την Πέμπτη θα αυξηθούν λογικά τα επιτόκια δανεισμού στην Ευρώπη στο 1,25%. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, αλλά επιδεινώνει την κατάσταση περαιτέρω. Αυτό, αυτή είναι η κατάσταση. 400 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε επενδύσει και έχουμε λύσει την κρίση. Σε καμία περίπτωση δεν την έχουμε λύσει. Αυτό που είναι απαραίτητο θεωρώ είναι μια προσέγγιση σε βάθος, την οποία δεν έχουμε επί του παρόντος. Να αναφερθώ στο Welling, στον πρόεδρο της, Ευρω... της ε, Ολλανδικής Τράπεζας, ο οποίος ε, δημοσίευσε την ετήσια έκθεση του ε, πρόσφατα και αναφέρει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες δεν είναι αρκετά αυστηροί. Αναφέρει ότι το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης είναι πολύ περιορισμένο. Το σύμφωνο για την Ευρώπη είναι πολύ αδύναμο γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός ε, υλοποίησης του. Και παραθέτω τον διοικητή της Εθνικής Ολλανδικής Τράπεζα, ο οποίος επαναλαμβάνει αυτά που είπαμε και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Τρίτο στοιχείο που αναφέρει ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος γίνεται υπερβολικά σε εθνικό επίπεδο και νομίζω ότι έχει δίκιο. Και μπορούμε να προσθέσουμε και κάποια στοιχεία μάλιστα. Πρώτο στοιχείο, το Ευρωπαϊκό Εκνοτικό Ταμείο. Τα προσωρινά και μόνιμα ε, ταμεία διάσωσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί προϋποθέτουν ομοφωνία αυτό δεν σημαίνει ότι όλη η Ευρωζώνη από εδώ και πέρα θα εκβιάζεται από τις ευρωσκεπτικές κυβερνήσεις και από τους πολιτικούς ε, αυτούς, εφόσον διατηρηθεί φυσικά αυτή η, αυτός ο κανόνα της ομοφωνίας. Και τέλος, και αυτό είναι το σημερινό μου μήνυμα, ε, δεν έχουμε ακόμα καθαρίσει το θέμα των ευρωπαϊκών τραπεζών. Το πρόβλημα δεν έχει ακόμη επιληθεί. Και η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη δεν πρόκειται να ξεκινήσει αν δεν αντιμετωπίσουμε πρώτα το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι μόνο το θέμα της οικονομικής κρίσης. Πλέον έχουν και ομόλογα στα χαρτοφυλάκια τους προβληματικών χωρών για τις οποίες οι αξιολογήσεις καταρακώνονται κάθε μέρα, κάθε βδομάδα. Εγώ τι ζητώ κύριε Μπαρόσο, εσείς και ο κύριος Τρίσε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να καταθέσετε το συντομότερο δυνατόν μια παγκόσμια καθολική συγγνώμη, αντίδραση στο πρόβλημα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται προ την κατεύθυνση αυτή και θέλουμε πραγματική οικονομική διακυβέρνηση γιατί υπάρχει αυτή η διακυβερνητική προσέγγιση χωρί κατάλληλου μηχανισμού. δεν πρόκειται να λειτουργήσει ούτε στο μέλλον όπω δεν λειτουργήσε και στο παρελθόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταθέσετε μία πρόταση και στα ταμεία διάσωση να καταργήσετε τον κανόνα ομοφωνία, γιατί έτσι δίνουμε δύναμη στις χώρες που είναι κατά του συστήματος και θα πρέπει να καταθέσετε ένα σχέδιο για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Δεν πρόκειται να ξεκινήσει η ανάκαμψη προτού προτείνεται έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό για να καθαρίσουν οι τράπεζες και όλοι ξέρουμε ότι θα χρειαστούν χρήματα για να επανα... επακεφαλοποιηθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες όπως είπε και ο κύριος Σούλτς προκειμένου να καλυφθούν και τα καλά, κακά δημοσιονομικά ε, κάποιων χωρών. Πού θα βρούμε τα χρήματα. Ο μοναδικός τρόπος να δημιουργηθούν αυτά τα χρήματα είναι να χρησιμοποιηθεί, να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ε, αγορά ομολόγων. Αυτή είναι η πραγματική λύση και θεωρώ κύριε Μπαρός ότι τελειώνει πια ο χρόνος. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε, θα πρέπει να σημειώσουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Χίφερ Χόφστατ, λέει ο Πρόεδρος και τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων ο Αντιπρόεδρος Ντανίλ Κον Μπέντιτ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς κύριε Βαν Ρομπόι, προς εσάς απευθυνθήκε ο κύριος Σούλτς και σας ανέφεραν γερμανικό τραγουδάκι. Όλα πάνε καλά είναι ο τίτλος στα γαλλικά, ουδέν πρόβλημα. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε τα πράγματα εδώ. Δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς. Αν μας αρέσει να σας ακούμε, διαβάζουμε και καμία εφημερίδα. Ξέρουμε τι τρέχει στο Συμβούλιο. Μη μας λέτε τώρα ιστοριούλε. Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα. Ε, δεν είμαστε εδώ για να χάνουμε το καιρό μας. Να σας πω κάτι. Και σε εσά και στον κύριο Μπαρόζο. Πάντα μιλάτε για σταθερότητα, για ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα. Ναι, πράγματι. Ξέρετε πώς ε, φτάνει το μήνυμα στους πολίτες πώς το πιάνουν. Ανισότητα, ε, αδικία, ε, ανασφάλεια. Έτσι το μεταφράζουν αυτοί. Και αν δεν αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορέσει να απαντήσει σε αυτά τα συναισθήματα περί αδικίας, περί ανισότητας, αυτό το συνέστημα της πραγματικότητας ανισότητας και το πρόσκαιρο της απασχόλησης, θα βλέπουν εκείνη την ανταγωνιστικότητα σαν κάτι που πέσει στο κεφάλι και στην πλάτη. Και εκεί έχουμε το πραγματικό πρόβλημα διότι οι μηχανισμοί διάσωσης των τραπεζών που θεωρώ ότι είναι πράγματι αναγκαίοι θεωρούνται από τους πολίτες όλα πάνε καλά για τις τράπεζες. Κοιτάτε τα κέρδη των τραπεζών. Κοιτάξτε τους μισθούς, τους παχυλούς. Μα λένε τρελοί, δαπανούν χρήματα και τα χρήματα τα πληρώσουν μετά οι πολίτες και οι εθνικοί προπολογισμοί. Ποιος θα τα πληρώσει και να αυξηθεί ακόμα παραπάνω η ανισότητα. Όλα τα στατιστικά στοιχεία τα τελευταία χρόνια μας δείχνουν ότι η ανισότητα αυξάνεται. Εάν δεν απαντήσουμε σε αυτό το πρόβλημα, οι πολίτες βλέπουν ένα κύμα, κύμα της άκρας δεξιάς, της αντιευρωπαϊστικής που αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το κύμα έχει ένα λόγο ύπαρξης. Είμαστε εμεί ανίκανοι να απαντήσουμε σε αυτά τα συναισθήματα περί ανισότητα, περί ε, και περί προσκέρου στην απασχόληση. Από τη στιγμή που δεν θα βρούμε απάντηση, θα τα καταφέρουμε. Ο Γκίβερ Χόφστα το είπε, ευρωομόλογα. Αυτό πρέπει να πούμε στους πολίτες και να τους κινητοποιήσουμε. Θέλουμε να υπάρχει ένα ταμείο υπεράσπισης άμυνας. Αλλά αν δεν υπάρχει ε, ταμείο επενδύσεων, αν δεν δείξουμε ακριβώς ότι θέλουμε να επαναπροωθήσουμε τον κινητήρα και χρειάζονται τα ευρωμόλογα. Όχι μόνο υπεράσπιση αλλά και επένδυση σε επενδύσεων. Εάν δεν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν οι πολίτες δεν θα καταλάβουν τίποτα. Δεν θα καταλάβουν αυτές τις πολιτικές και πρέπει να λέμε τα πράγματα από το όνομά τους. Ανισότητα. Γιατί δεν είναι δυνατόν σήμερα να ληφθούν κάποια κοινωνικά μέτρα στην Ευρώπη. Να τα συζητούν οι πολίτες. Να αποφασίσουμε έναν ελάχιστο μισθό, Φερρυπίν, για όλη την Ευρώπη. Ε, ένα ιδέα ενό ελάχιστου μισθού, όχι στο ίδιο επίπεδο. Είναι απίστευτο μια χώρα όπω η Γερμανία ε, ε, να, προσπαθεί να εξισορροπήσει οικονομικά, να μην συζητά αυτό το θέμα. Και είναι από τι λίγε χώρε που είναι κερδοφόρε στην Ευρώπη σήμερα η Γερμανία και δεν μπορεί να εγκαθιδρύσει έναν ελάχιστο μισθό για του πολίτε τη. Είναι κάτι που πρέπει να τεθεί στο θέμα αυτό τη οικονομική και κοινωνική κυβερνήσεω τη Ευρώπη για τη Λιβύη. Σωστά τα είπε ο Μάρτιν Σούλτ. Είναι δραματική η κατάσταση. Είναι μια χώρα όπως η Γερμανία που κρύβεται και άλλες χώρες που προσπάθησαν να ανταποκριθούν και να απαντήσουν και πρέπει να πω και συμφωνώ. Πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό που θα ήθελα όμως όταν συζητάμε για μια πολιτική γειτονία να κάνουμε απολογισμό των ανοησιών που κάναμε πριν στην πολιτική της γειτονίας. Τη σχέση με τον κύριο Γκαντάφη πριν. Τι κάναμε πριν το βομβαρδίσουμε. Ποιες ήταν οι σχέσεις των ευρωπαϊκών χωρών με τον κύριο Γκαντάφη, με τον κύριο Μπεναλή, με τον κύριο Μουμπάρακ. Ας κάνουμε επιτέλους έναν απολογισμό αυτό που περιλαμβάνονται συμφωνίες σύνδεσης. Τα άρθρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πόσο μετράνε για μας. Νάδα. Τίποτα. Μηδέν. Εάν δεν κάνουμε λοιπόν την αξιολόγηση, ας σταματήσουμε να ψευδόμεθα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, έδωσε πέντε λεπτά για να το σκεφτεί. Τι δεν κάναμε πριν ε, ασκήσουμε την πολιτική της Μεσογείου. Το σκεφτήκατε. Εγώ δεν διάβασα τίποτα σε εφημερίδες. Τίποτα δεν άκουσα από αυτά που είπατε πάνω σε αυτό. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν ικανό να δείξει ελάχιστη, να κάνει ελάχιστη αυτοκριτική. Ελάχιστη αυτοκριτική του τι δεν κάναμε πριν, τι δεν κάναν πριν για την Ιαπωνία τώρα. Το πρόβλημα το, για μεγαλύτερη πυρηνική ασφάλεια είναι να φύγουμε από την πυρηνική ασφάλεια. Δεν υπάρχει μηδενική, μηδενικός κίνδυνος στον πυρηνικό τομέα. Δεν μπορεί εν μία ανοιχτή να το πετύχουμε. Αν δεν βγούμε από την πυρηνική ενέργεια θα υπάρξει ασφάλεια. Και το πρόβλημα δεν είναι δοκιμές αντοχής. Ένα τύχημα. Το πρόβλημα είναι ο κ. Δακώστο, ο οποίο είναι πρόεδρο τη Υπηρεσία Ασφαλεία τη Πυρηνική τη Γαλλία, είπε το απίστευτο. Μέχρι τώρα ποτέ δεν μελετήσαμε την σόρευση δυνατοτήτων, πιθανοτήτων για το ατύχημα. Αυτό είναι η Ιαπωνία. Δεν είναι ένα ατύχημα. Είναι συσσόρευση 4-5 ατυχημάτων συν ανθρώπινα σφάλματα που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Είναι αδύνατον μαθηματικός να εξασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια. Όσο οι Ευρωπαίοι δεν το κάνουν αυτό, δεν θα βγούμε μια νυχτή, αλλά αν δεν βγούμε από την πυρηνική ενέργεια, σταματήσουμε να μιλάμε για ασφάλεια. Ασφάλεια απόλυτη δεν υπάρχει στον πυρηνικό τομέα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για, από τους ειδικού και μεταρρυθμιστές ο κ. Ζαχραντήλ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Το πιο σημαντικό που αναφέρθηκε θέμα στη Συμβούλιο ήταν η οικονομία, η σταθερότητα της Ευρωζώνης, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην ομάδα μας οι περισσότεροι βουλευτές είναι από χώρε που δεν είναι στην Ευρωζώνη και η πλειοψηφία των βουλευτών έρχεται από χώρε που δεν είναι στο σύμφωνο για το ευρώ. Ε, δεν θέλουμε να αποτύχει το ευρώ όμως βέβαια. Θέλουμε μια Ευρώπη που να ζει στην ευμάρεια. Θέλουμε κυβερνήσεις υπεύθυνε που θα σταματήσουν το πρόβλημα της ε, χρέωσης του δημόσιου τομέα που θα κάνουν τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται και θα λάβουν μέτρα που θα οδηγήσουν στην ε, αποκατάσταση πειθαρχίας της χρηματοπιστωτικής. Όλα αυτά είναι σωστά. Αυτό που είναι άδικο και αυτό που μας ενοχλεί είναι το κρυφό πρόγραμμα κάποιων κρατών μελών και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρυφό πρόγραμμα κάποιων πολιτικών ομάδων που προσπαθούν να το περάσουν. Εκμετάλλευση δηλαδή της κρίσης για νέα μετακίνηση των αρμοδιοτήτων, να προχωρήσει φορολογική εναρμόνιση, να πάμε προς φορολογική ένωση και ένα νέο βήμα προς την πολιτική ολοκλήρωση. Εμείς λέμε όχι σε αυτή την ένωση, δεν θέλουμε τέτοιου είδου ένωση. Είμαι εδώ από το 2004 και κάθε φορά που υπάρχουν δυσκολίε ακούω μία μονοφράση. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη. Λένε, χρειάζεται περισσότερο κοινοτική μέθοδο. Εγώ λέω όχι, δεν χρειαζόμαστε όλα αυτά, δεν τα χρειαζόμαστε. Ε, οι προσπάθειε να επιλύσουμε τα πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μα οδήγησαν στην κατάσταση τώρα από την οποία προσπαθούμε να βγούμε. Πρέπει να καταλάβετε επιτέλου ότι Έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σταματήστε να ζείτε 50 χρόνια στο παρελθόν. Το ευρωπαϊκό παράδειγμα άλλαξε, το πρότυπο άλλαξε και καλό θα ήταν να μην επιμένετε από αυτού. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο Λόταρ Μπίσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της, ε, του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της ε, Επιτροπής. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα δεν είναι επαρκή του Συμβουλίου. Καταρχάς, ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική. Αυτά που βλέπουμε, ε, σας είπαμε μάλλον, ε, και εκφράσαμε σε ακρόαση τι θεωρούμε για τα οικονομικά μέτρα. Αυτό που θέλουμε είναι να ξεπεράσουμε τα νεοφιλελεύθερα κερδοσκοπικά μέτρα και σε ό,τι αφορά μέτρα όπως το Flex Security. Αυτό που είναι απαραίτητο θεωρούμε είναι η δημοκρατική νομιμοποίηση και ο έλεγχος της ε, οικονομικής πολιτικής και, και η φορολογία για το dumping σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα πρότυπα που επιβάλλονται. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών προκειμένου να ε, αποφευθούν και κίνδυνοι που ελοχεύουν. Σε ό,τι αφορά την Λιβύη, στην Βόρειο Αφρική, κυρίως στη Λιβύη, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν σε μια μακάβρια κατάσταση. Πολλά ακούσαμε από τους συναδέλφους ως κριτική. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Ο δικτάτορας Καντάφη καταπολεμάει τους ε, διαμαρτυρόμενους ε, και τους άμαχους με τα όπλα που αγόρασε από εμά. Το πυροβολούν τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ και οι αγωνιστές για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη οι οποίοι επίσης χρησιμοποιούν όπλα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποιος είναι ο κώδικας κατά της εμπορίας όπλων που επιτρέπει μια τέτοια κατάσταση. Πού είναι η υποστήριξη της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του αγώνα κατά των κοινωνικών αδικιών όταν στην Λαπεντούζα ε, κάθε μέρα είναι εκατοντάδες οι πρόσφυγες από τη Βόρεια Αφρική. Φοβάμαι ότι και σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα που προτείνεται για την γειτονία, το μόνο που προωθούμε είναι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Δεν εστιάζουμε στις ανάγκες των χωρών εταίρων. Κατά τρίτον, η Ιαπωνία. Σήμερα το απόγευμα και αύριο έχουμε χρόνο συζήτησης για την Ιαπωνία και στο σημείο αυτό Χρειάζεται μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση η οποία δεν υπάρχει σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτά τα επωνομαζόμενα stress στην την πολιτική ασφάλειας. Δεν μου προκαλεί έκπληξη ο σκεπτικισμός των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναρωτιούνται τι ακριβώς αντιπροσωπεύει πια αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Gottfried Bloom από την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Well, είναι ενδιαφέρον. με επιτρέπετε, θα ήθελα να μιλήσω για τη Λιβύη. Πότε κατάλαβαν οι μεγάλοι και οι καλοί ότι είναι κακός ο Καντάφη, πια, μετά από την φωτογράφηση που και εσείς τον εναγκαλιζώσετε κύριε Πρόεδρε, πότε ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος είναι κακός. Γιατί πρέπει να σας πω ότι τα θύματα του Λόκερμπι στη Σκωτία και τα θύματα των αποτροπιαστικών ενεργειών του Ήρα γνωρίζανε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Όμως ο Γκαντάφη έχει χρήμα και έχει πετρέλαιο και έτσι όλοι κλείνετε τα μάτια, έτσι δεν ήταν. Να όμως που όμως γύρισε μπούμεραγκ το ρόλο αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι το χειρότερο είναι ε, ο Πρωθυπουργό ε, της Βρετανίας, ε, ο οποίος αφού έχει και τις ενόπλες δυνάμεις, στο βασιλικό ναυτικό, τελείως καταστρέψει, λέει τώρα ότι είναι συντα... συντηρητικός. Και ξέρω επίσης ότι μιλάμε πολύ για τη βία κατά πολιτών, μιλάμε για τη δημοκρατία. Στη Ζιμπάμπου έχουμε αυτόν τον, τον, τον άνθρωπο εκεί πέρα που δεν μας ενδιαφέρει αυτά που κάνει γιατί δεν έχει χρήματα και δεν έχει πετρέλαιο. Δεν είμαστε υποκριτές. Ε, Ευχαριστώ. Μπάρι Μάντλενερ από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Μπαρόσο, σας ε, κάνουμε το κέφι. Θα υπάρχει για το ευρώ ένα μόνιμο μηχανισμό διάσωσης, ε, ένα ταμείο για τις χώρες οι οποίες ε, έκαναν, τα πήγαν πάρα πολύ άσχημα, που, που τις ενταμείω αυτές τις χώρες και που τιμωρεί τις χώρες που ακολούθησαν δημοσιονομική πειθαρχία. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία δίνει καλά δάνεια στις χώρες εκείνες οι οποίες εξαπάτησαν το Ταμείο. Και πού πάνε τα χρήματα αυτά. Συμμετέχουν όλες οι χώρες και η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Οι χώρες όμως αυτές δεν έχουν ε, λεφτά. Άρα τι σημαίνει αυτό κύριε Πρόεδρε. Οι χώρες που τα πήγαν καλά, η Ολλανδία θα πληρώσουν. Οι Ολλανδοί πολίτες θα πληρώσουν τα χρέη της Ελλάδας, της Πορτογαλίας από που προέρχεστε κι εσεί, κύριε Μπαρόσο και αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο, δεν είναι αλληλεγγύη αυτό. Αυτό ανταμείβει την κακή συμπεριφορά κάποιων ε, ε κακών χωρών και αυτό εις βάρος ε, των τίμιων εργαζομένων ε, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Θα πρέπει να να εκδιωχθούν αυτές οι χώρες από την Ευρωζώνη, να ξαναεισάγει η Ελλάδα την δραχμή και η Πορτοκαλία το Εσκούδο και να αποκλειστούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Ο κύριος Βέρνερ Λάγκε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι ένα σημαντικό ενδιάμεσο βήμα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον αν συνεχιστούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθερότητας ε, και συνεχίσει η κατάσταση όσο έχει, το χαρτί αυτό δεν αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν δεν συμφωνώ με την αισιοδοξία των δύο προέδρων ότι αντιπαρήλθαμε πλέον την κρίση. Όχι, θα κρυθούν αυτά στο μέλλον. Έχουμε δυόμιση χρόνια μετά από την πτώχευση της Λέμαν. Και πού βρισκόμαστε ο αρμόδιος ε, ε, Επίτροπος απέριψε τις ε, προτάσεις για τη φορολογία. Θέλω πλέον αποτελέσματα, γιατί το, το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία ε, πρόωθησε 12 αποφάσεις σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, τις οποίες αρνήθηκε ο τότε Επίτροπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήθελε λοιπόν να προωθήσει την επίλυση των προβλημάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, διαπιστώσαμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους εθνικούς ε, εγωισμούς και θα πρέπει να ενδυναμωθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν λοιπόν λόγοι για αισιοδοξία και θα πρέπει να δικαιώσουν τον κύριο Φερχόφστατ. Η ενίσχυση του προπολογισμού δεν είναι επαρκής. Η διακυβέρνηση δεν είναι δεσμευτική και εξακολουθούν να υπερισχύουν τα εθνικά συμφέροντα. Αν δεν έχουμε λοιπόν την τόλμη, την τόλμη για περισσότερη Ευρώπη η οποία θα πρέπει να απαιτηθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις δεν θα υπάρξουν διαρκείς και βιώσιμες ε, λύσεις. Κύριε Μπαρόσο, οι Έλληνες συνάδελφοι καταψήφισαν το πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν συμφωνώ με τον ε, κύριο Σούλτς ουσιαστικά αλλά στην περίπτωση της Πορτογαλίας και το δικό σας κόμμα καταψήφισε το πρόγραμμα αυτό. Και αυτό δεν επιτρέπεται να συμβαίνει στην Ευρώπη. Να παρακαλέσω όλους λοιπόν να βοηθήσουν αυτό το πρόγραμμα εθνικών ε, λύσεων να μην έχει μέλλον. Ähm, Ευχαριστώ. Η κυρία Εστρέλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχει ένα θέμα, ερώτημα που θέτουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Το, οι αποφάσει του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μας βοηθήσουν να βγούμε από την κρίση. Αυτό διερωτώνται οι πολίτες. Πολλοί ίσως να θεωρούν ότι αυτές οι αποφάσεις ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Όμως δεν είναι αρκετά φιλόδοξες. Αυτό πιστεύουν. Αυτοί που είδαν, αυτοί που βλέπουν τα διάφορα έγγραφα Εάν έβλεπαν τις εσωτερικές διεργασίες ίσως να θεωρούσαν ότι κινούνται κάποιοι με κερδοσκοπικούς στόχους και θα διερωτώνται τι κάνει η Ευρώπη για να δημιουργηθούν φορείς βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που να είναι αξιόπιστοι ε, και υπόθηκε ότι θα πρέπει, αν κάποια χώρα μπορεί να βρει μια λύση να βγει από την κρίση μόνη να το κάνει, γιατί είναι πολύ δαπανηρό πάρει δάνεια. Το ίδιο θεωρεί και η Πορτογαλία. Χρειάζεται χρηματοδότηση η οικονομία της Πορτογαλίας και χρειάζεται επίσης η Πορτογαλία λογικά επιτόκια. Αλλά οι φορείς βαθμολόγηση επιστοληπτικής ικανότητας είναι βορρά των ε, κερδοσκόπων και τελικά ε, βγάζουν χρήματα οι κερδοσκόποι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη τελικά που αποδίδεται στην Ευρώπη. Εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια κρίση της Ευρωζώνης που περνάμε. Αυτές οι επιθέσεις επί του κρατικού χρέους έχουν σαν στόχο την υπονόμευση του ευρώ, του ενίου νομίσματος και του ευρωπαϊκού προγράμματος εν γέννη, του οικοδομήματος. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτεί μια ευρωπαϊκή απάντηση. Αν θέλουμε να φύγουμε από την Ευρώπη, χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε να πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις τωρινές και τις μελλοντικέ βάσει της εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε από την παραδούσα απορία μας. Θα πρέπει ε, να μας υποστηρίξουν πολίτες. Χωρίς τους πολίτες δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Γκουλάρ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ε, μας ε, ζωγραφίσατε ένα θετικό, θετική εικόνα των συζητήσεων. Υπάρχουν θετικά στοιχεία, δεν θα αναφερθώ ξανά σε αυτά. Έχω κάποια ανησυχία όμω, η οποία ξεπερνά τις τεχνικές λεπτομέρειες και αυτά που μας είπατε. Είναι η διαφορά βορρά-νότου που δημιουργείται, η ρογμή βορρά-νότου. Ακούμε κάποιους που λένε ότι έχουν δίκιο η μεν και άδικο η δε, η μεν είναι καλή, η δε είναι κακή και φαίνεται την αλληλοεξάρτηση που υπάρχει. Και αυτό είναι σοβαρό. Και στην άρνηση αντιμετωπίσεως του προβλήματος των τραπεζών που ανέφερε ο κ. Βαν εκεί υπάρχει άρνηση σε κάποιες χώρες του Βορρά που δίνουν μαθήματα στον Νότο να δουν αυτές ποιες ευθύνε έχουν. Πιστεύω ότι αν ένα καθήκον είναι στα χέρια μας κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κύριε Μπαρόσο είναι να αποφύγουμε πάση θυσία να παραταθεί και να δρεωθεί αυτή η διαφορά, αυτή η ρογμή. χρειάζονται λύσεις που καλύπτουν όλους. Όλοι πρέπει να υπομιστούν τις ευθύνες τους. Και τέλος, βρίσκονται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι εξαιρετικά, ασχολείται ομφαλοσκοπή. Όλες οι συζητήσεις γίνονται σαν το ευρώ να μην έχει στόχους παγκόσμιας εμβέλειας. Δεν υπάρχει τίποτα ε, όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση του ευρώ στο Εθνικό Νομισματικό Ταμείο. Η Γαλλία που έχει την προεδρία του z 20 θέλει να κάνει νομισματική μεταρρύθμιση σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν υπάρχουν προτάσει όπω αυτή των ευρωμολόγων που θέλουμε να προωθήσουμε που έχουν σαν στόχο να κάνουν το ευρώ πραγματικά ένα παγκόσμιο νόμισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαμπέρ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Σέβομαι και το πρόσωπό σας ε, και το έργο που επιτελείτε. Δεν με πείσατε πάντως. Λέτε ότι δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι να ανησυχούν γιατί εμείς δουλεύουμε για αυτούς. Εγώ αυτό που διαβάζω όταν βλέπω αυτό το, αυτή τη δέσμη ε, EuroSyn, όταν λέμε ανταγωνιστικότητα, τι εννοούμε, να μειώσουμε τους περικοπούς, ε, τις περικοπές, λιγότερη ασφάλεια, περισσότερη ευελιξία Τίποτα δεν λέμε για την παραγωγικότητα σε ό,τι αφορά τους σπόρους ή σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Εγώ θα σας πω το εξή. Ποτέ δεν θα μετωπίσουμε την Κίνα σε ό,τι αφορά ε, τους μισθούς. Η Κίνα θα μας κερδίσει και σε ό,τι αφορά τους σπόρους και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Μα πού πηγαίνουμε τελικά, τι μένει για την Ευρώπη. Λέτε ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για κοινωνικά επιδόματα έχουμε κάποιου στόχου λογικού. Λέτε όμω πρέπει να μειώσουμε τι δαπάνε. Το 40% των δαπανών είναι κοινωνικέ. Λέτε να μην ανησυχούμε. Άμα περισταλούν, να μην ανησυχούμε. Λέτε ε, μην ανησυχούμε, έχουμε τα έσοδα. Έχουμε την ε, βάση φορολογίας για τις επιχειρήσεις. Μα είναι αστείο αυτό που προτείνετε. Μιλάτε στην ευκτική. Λέτε ότι θα είναι αυτή η άποψή μας και θα κάνουμε αυτά σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Μα οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν. Εγώ δεν έχω δει ποτέ σε ό,τι αφορά τις φορολογικές επιλογές κανέναν να επιλέγει αυτό που θα του στοιχήσει περισσότερο. Ποιος δεν πρέπει να ανησυχεί. Μόνο η μέτοχοι των τραπεζών. Μας μιλάτε για δοκιμές αντοχής. Αυτό που έγινε πέρυσι ήταν φάρσα. Ε, ίσως κακή φάρσα να είναι και αυτό που θα κάνετε φέτος. Ακόμη και είναι σοβαρές αυτές οι δοκιμές αντοχής. Τελικά ποιος θα δώσει Ποιο θα επανακεφαλοποιήσει τι τράπεζε, εμεί. Τελικά, το ιδιωτικό κεφάλαιο, πώ να μην ανησυχούμε. Και τέλο, δεν μιλάμε για τον ελέφαντα που είναι στο σαλόνι μας, το Ιρλανδικό και το ελληνικό χρέος. Ξέρετε πολύ καλά ότι όπως και να το δούμε δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν ε, το, τα ποσά που θα τους δώσουμε. Και ποτέ δεν θα είναι εύκολο το εγχείρημα αυτό και το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό μας κοστίσει πολύ ακριβά. Ευχαριστώ. Επόμενος ο κύριος Κάλεμαν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, συχνά πέφτει στην παγίδα να χρησιμοποιήσει γραφειοκρατικές λύσεις οι οποίες δεν είναι αναλογικές στη σοβαρότητα του προβλήματος. Το ίδιο σφάλμα κάνουμε τώρα σε ό,τι αφορά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση. Είναι σοβαρή και προαπαιτεί την ανάληψη δράσης, αλλά πολλές από τις προτινόμενες ε, ε, λύσεις θα μας ζημιώσουν μακροπρόθεσμα στο μέλλον χρησιμοποιείται η ευκαιρία από πολλούς να ξεκινήσουν σχέδια οικονομικής διακυβέρνησης με παρέμβαση και έλεγχο ως αρχές προσανατολισμού. Οι λύσεις που προτείνονται είναι καταρχάς να καταχραστούμε του εφιστάμενους κανόνες όπως το άρθρο 1-2-2 για τις συνθήκες που ποτέ δεν είχε ως σκοπό τέτοιες διασώσεις για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε και θεωρώ ότι θα αμφισβητηθεί στο Ευρωπαϊκό ε, Δικαστήριο και θα επιβάλλει πιο πολλού περιορισμού στα κράτη-μέλη, θα περιορίσει δηλαδή τι δημοκρατικέ επιλογέ του εκλογικού σώματο. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ιρλανδία. Έκανε ό,τι μπορούσε για να σταθεροποιήσει το τραπεζικό κλάδο, μια σταθεροποίηση η οποία χρειάζεται για τις τράπεζες και τους θεσμούς και άλλων κρατών μέλων παρεπιπτόντος που ιδάλλως θα είχαν τεράστια έκθεση και ανταμείβονται με ε, τις αξιώσεις ε, των άλλων κρατών μελών για να αυξηθούν τα επιτόκια συνεργασίας, το οποίο είναι και μη δημοκρατικό και πραγματικά άδικο, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Ντεμπρίν για ένα λεπτό. Uh, Τι είδου σκέψεις προσανατολίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και τους κάνουν να πιστεύουν ότι οι περιορισμοί που ετέθησαν επί της Ιρλανδίας δεν θα αυξήσουν το χρέος. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα αν εφαρμοστούν οι πολιτικές που μας προτείνουν. Να αυξηθεί το χρέος μας. Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών που συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής για περιορισμούς ε, οικονομικούς ε, που περιορίζουν και την ευμάρεια των ε, ανθρώπων. Περικοπές. Ε, μείωση των δυνατοτήτων των κρατών μελών να μπορούν να οδηγηθούν προς την ανάπτυξη. Αυτά επευλήθησαν, τέτοια μέτρα επευλήθησαν στην Ιρλανδία. Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ε, αυστηρές περικοπές. Τι σημαίνει αυτό, απώλεια θέσεων εργασίας, σοβαρή μείωση της παροχής δημοσίων υπηρεσιών. Το βάρος του Ιρλανδικού χρέους δεν μπορεί να το σηκώσει η Ιρλανδία αν κάποιο από το βάρος ε, δεν το πάρουν κάποιοι ε, οι τράπεζες, τότε θα αποτύχει, θα η Ιρλανδία. Η κυρία Τζαβέλα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Σύμφωνο για την Ευρωπαϊκή Σταθερότητα έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Πώς μπορούμε να πετύχουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην οικονομία όταν η εργασιακή αγορά τη χάνει κατάχρασης από την νόμιμη μετανάστευση και όταν τα ευρωπαϊκά προϊόντα αντικαθεστούνται από προϊόντα τα οποία εισάγονται από χώρες της Ανατολής όπου υπάρχει έντοση εργασίας. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να προστατεύσουμε τα γεωγραφικά μας και οικονομικά μας προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο πιο καλά το κάνουμε αυτό, τόσο το καλύτερο για μας, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η πρότασή μου είναι να ενσωματώσουμε τα συστήματα ταυτοποίησης ε, και προστασία των οικονομικών και γεωγραφικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Ιδάλλως δεν θα πετύχουμε την ανταγωνιστική Ευρώπη που θέλουμε μέσα σε ένα πολύ εχθρικό οικονομικό περιβάλλον το οποίο επικρατεί παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα ο κύριος Φανχέκε για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε όταν η κρίση, αν μας δείχνει κάτι η κρίση στη Λιβύη, είναι καταρχάς την έλλειψη σοβαρής ε, γεωπολιτικής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Είναι η λυπηρή πραγματικότητα ότι η παρέμβασή μας εκεί αποτελεί απόρρια καταρχάς μιας ενιαίας ε, εσωτερικής πολιτικής του Σαρκοζή. Συγκυριακής είναι επίσης περίεργο το γεγονός ότι όλοι στο ημισφαίριο αυτό, οι οποίοι ενίστανται και δικαίως κατά του καθεστώτος του Καντάφη, μέχρι πρόσφατα με μεγάλα χαμόγελα φωτογραφούνταν δίπλα του και τον υποδέχονταν με στρατιωτικές τιμές. Είναι πιο απλό σήμερα να πυροβολούμε τον Καντάφη παρά να δίνουμε απαντήσεις στα τεράστια ερωτήματα που ανακύπτουν. Να αναφέρω ένα. Οι επαναστάτες οι οποίοι είναι ετερογενείς ως ομάδα και μερικοί εξ αυτών είναι, αν θέλετε, πνευματικά στο μεσαίωνα. Θα τους υποδεχτούμε και τι εγγύηση έχουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα όπλα που υπάρχουν για να βυθιστεί η χώρα σε μεγαλύτερη κρίση. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πιο μεγάλη παρουσία στην προστασία την στρατιωτική των εξωτερικών μας συνόρων γιατί εκεί υπάρχει ένας τρομακτικός πόλεμος τον οποίο δεν ε, συζητάει κανένας και εκεί χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα και ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος η κυρία Βόρτμαν Κόλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε. Το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ελήφθησαν αποφάσεις οι οποίες ήταν πραγματικά διανόητες πριν από ένα χρόνο και θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ και τον Πρόεδρο Φανρόμπα και τον ε, Πρόεδρο Μπαρόσο. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αλλά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο δρόμο που έχουμε να διανύσουμε για να ε, ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη στην οικονομία μας και στο, στην Ευρωζώνη, για να βγούμε από την κρίση με οικονομική ε, ανάπτυξη. Το κοινοβούλιο αυτό έχει ρόλο συναπόφαση, συνομοθέτη σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Και εδώ θέλουμε πιο πολύ φιλοδοξία. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστούν οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από πλευράς μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, πιο ε, ισχυρή εποπτεία που θα βασιστεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσατε διάφορους συναδέλφους οι οποίοι ανέφεραν ότι θέλουν μια αντίστροφη διαδικασία ψηφοφορίας και ότι θέλουν πολύ πιο ε, καλό κοινωνικό συντονισμό και αυτό ξεπερνάει τις δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη στρατηγική του 2020 αναφέρονται οι αρχές της κοινωνικής αγοράς που ε, θέλουμε προκειμένου να πετύχουμε τις θέσεις απασχόλησης, να προωθήσουμε τις θέσεις απασχόλησης και την ανάπτυξη. Τους στόχους αυτούς, άκουσα να το αναφέρει αυτό και ο πρόεδρος Μπαρόσο, θέλουμε να εξασφαλιστούν σε ό,τι αφορά τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και θα καταθέσουμε σχετικές προτάσεις. Τονίζεται ότι θέλετε τον Ιούνιο να έχει επιτευχθεί μία συμφωνία σε ό,τι αφορά την προτάση αυτή. Μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε να προωθείτε τις προτάσεις αυτές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί μόνο έτσι θα πετύχουμε συμφωνία τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Βόρτμαν Κόλ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ντερόσα για δύο λεπτά. Thank you very much, uh, Madam. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε να ρωτήσω κάποιε ειλικρινεί ερωτήσεις απευθυνόμενο ε, προς την Τρόικα, στην το Συμβούλιο του Ευρωπαίου φορεί. Σοβαρά λέτε ότι θέλετε να σώσετε την Ευρωζώνη και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα το οικοδόμημα. Οι δοκιμέ αντοχή των τραπεζών ολοκληρώθηκαν και κατέληξαν στα πιο απεσιόδεξα σενάρια για την Ιρλανδία. Η κυβέρνησή μας ε, τελικά την κόκκινη γραμμή στον αφάσι τράπεζε αποφάσεις ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές όσον αφορά τους μεγάλους μετόχους ε, της ε, ε, Τράπεζας Ιρλανδίας και της Allied Irish Bank. Γιατί δεν κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά την ενδιάμεση χρηματοδότηση, τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση των τραπεζών. Γιατί ο κ. Σαρκοζή και η κυρία Μέρκελ επιμένουν επί τη καταστροφή τη Ιρλανδική βιομηχανική βάσεω σε αντάλλαγμα διάσωση τη οικονομία Ιρλανδίας. Γιατί κάποια κράτη-μέλη μπλοκάρουν την πρόοδο όσον αφορά τον φόρο επί τον, Ευρω... τον ευρωπαϊκό επί των χρησιμοποιητικών συναλλαγών και για τα ευρωμόλογα. Γιατί έχουμε περικοπές του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Σύντομη απάντηση. Υπολογισμοί εκλογικοί, βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και δογματικά οικονομικά. Η κρίση της Ιρλανδίας είναι ένα απόσπαστο τμήμα της κρίσης της Ευρώπης. Η αποτυχία της Ιρλανδικής οικονομίας δεν θα είναι μόνο αποτυχία για την Ευρώπη, αλλά και της αποτυχία της Ευρώπης. Λοιπόν, ε, είναι κρίσιμο το πρόβλημα τη Ιρλανδία, το χρέο. Και το κουαρτέτο θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό σε αυτή την επίλυση του θέματο. Τι θέλουμε από το κουαρτέτο, φαντασία, όραμα στι διαπραγματεύσει με την Ιρλανδία. Και σημειώστε αυτά που λέω τώρα, έτσι. Η Ιρλανδία είναι δημοκρατία. Όπω η Γαλλία, όπω η Γερμανία, όπω η Φιλανδία. Κυβερνούμε βάσει τη ε, βουλήσεω του λαού. Το εκλογικό σώμα τη Ιρλανδία δέχτηκε σοβαρά μέτρα λιτότητα Θέλει να σφίξει τα δόντια να πνίξει το θυμό του, αλλά θέλει δίκαιου όρου από πλευρά Ευρώπη. Αλλιώ η αντοχή, η ανοχή ε, τελικά θα εκραγεί, θα πάψει η ανοχή πλευρά και του λαού και τη κυβερνήσεω. Ευχαριστώ και τώρα δούμε στον κύριο Χάκλοντ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω πάνω σε μια θετική νότα. Και πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ στις ανησυχίες που εκφράστηκαν μόλις τώρα. Υπάρχει κάτι θετικό ότι τελικά φτάσαμε στην διακυβέρνηση τη μακροοικονομική και σχετικά μέτρα. Ο Ιρλανδός συνάδελφος μας υπενθύμησε τις ανησυχίες του μόλις τώρα. Αλλά σίγουρα στο μέλλον θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και επί μακροοικονομικών πτυχών. Πιστεύω ότι αυτά που γίνονται τώρα είναι σημαντική πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει ανάγκη αλλαγής, πράγματι. Αλλαγής όσον αφορά τη διακυβέρνηση, το governance. Να μην επικρατεί πάντα μόνο το εμπορικό πνεύμα. Να μην γίνονται συνεχώς παζαρέματα. Κυρίως όταν λαμβάνονται αποφάσεις στο Συμβούλιο. Όμως οι αποφάσεις που ελήφθησαν, ελήφθησαν βάσει συστάσεων. Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποια τάση στο Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποιες τάσεις στο Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις όπως της Φινλανδίας στο Συμβούλιο. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Λυπούμε δεν σημαίνει ότι όλη η Φιλανδία υποστηρίζει την τοποθέτηση που ακολουθείται. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Έφνερ. Δεν τον βλέπω όμως στην αίθουσα. Dann hat jetzt das Wort Herr für... δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σιμάνσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η νέα χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην προσπάθεια ενίσχυσης κανόνων ε, για την περιστολή των δαπανών που είναι υγιείς κανόνες αλλά μη υγιείς κανόνες για την ε, μείωση της εθνικής ε, και φορολογικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Αμφιβάλλω λοιπόν τα μάλλα ότι οι χώρες του Europlus, του Eurosyn θα μπορέσουν να επιβάλλουν αυτά τα μέτρα συλλογικά εάν δεν μπορούν να το κάνουν ατομικά. Τώρα, η ενοποίηση, η παγίωση φορολογική βάση είναι ένα καλό μέτρο προ ε, την ε, φορολογική ένωση που στόχο έχει μόνο την κατάργηση, την εξάλληψη του φορολογικού ανταγωνισμού. Η Λαγκάρντ, ο Σαρκοζή πριν από τέσσερι ε, μήνε επέμεναν να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστέ στην Ιρλανδία με πρόσχημα την καταπολέμηση τη κρίση. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών πάντως είναι μια συνταγή για να παραμείνει η κρίση και όχι για να μετριαστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τους συναδέλφους που ζητούν το λόγο για την διαδικασία Catch the Eye. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ήδη 20 άτομα που έχουν ε, ζητήσει το λόγο και δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο ε, πριν από την ψηφοφορία. Ωστόσο, μπορείτε να ζητάτε το λόγο παρόλα αυτά. Ο κύριος Μέρφυ έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Στις 19 Ιανουαρίου, απαντώντας στον Τζον Χίγγινς, είπατε κύριε Μπαρόσο σε αυτή την αίθουσα ότι η Ευρώπη προσπαθεί να υποστηρίξει την Ιρλανδία. Με την... το Φίνα η κυβέρνηση εργατικής Φίνα υποχώρησε στους συμφέροντα των μετόχων και έτσι ούτε το Συμβόλαιο ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουν. Αλλά εργατική τάξη στην Ιρλανδία και στην Ευρώπη είναι που υποχρεώνονται να υποστηρίξουν τι ευρωπαϊκέ τράπεζε και του κερδοσκόπου πληρώνοντα τι απώλειέ του. Οι προτάσει για οικονομική διακυβέρνηση αντιπροσωπεύουν αυτή την απόπειρα να παγιωθούν οι περικοπέ των μισθών περικοπέ. Η βαθμολόγηση τη λιτότητα, εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ περικοπών εξασφαλίζουν ότι παρά τι αντιρρήσει του οι εργαζόμενοι πληρώνουν τελικά για την κρίση. Αυτό το, αυτό δόγμα σοκ της Ευρώπης ε, προσπαθούν να βγάλουν μέτρα και να αποφύγουν δημοψηφίσματα. Η αριστερά στην Ιρλανδία θα πετήσει δημοψήφισμα για την πρόταση για μόνιμη λιτότητα που προσπαθεί να επιβληθεί. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Ρώση για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Αξιότιμοι συνάδελφοι, αυτό το Συμβούλιο αναφέρθηκε σε τρία σημαντικά θέματα. Την καταστροφή του περιβάλλοντο στην Ιαπωνία με το περιβηνικό ατύχημα, η κρηματοπιστική κρίση για την Ευρώπη και η κατάσταση στο Μαγκρέμπ. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, παρόλο που είμαστε πολύ κοντά στο λαό που επλήγει τόσο σκληρά, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την αναθόρηση των εμπορικών συμφωνιών ει βάρο των επιχειρήσεων μα. Αντίθετα, είμαστε υπέρ παρέμβαση με μέσα ανθρώπου και χρήματα, ανθρωπιστική βοήθεια. Όσον αφορά με τη ειδική κρίση, ε, είναι ουτοπικό να πούμε ότι πέρασε. Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει ένα πακέτο παρεμβάσεων για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βγουν από την παρούσα κατάσταση, να εξασφαλίζονται σταθερότητα σε όλη την Ευρωζώνη. Είμαστε υπέρ επίση και τη μειώσεω του βάρου ε, τη νομοθεσία και τη γραφειοκρατία και να προωθήσουμε ανταλλαγέ με τρίτε χώρε με τον όλο ότι θα είναι αμοιβαία τα ωφέλη. Όσον αφορά το Μαγκρέ, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε, είχε πάρα πολύ κακή εικόνα που προέβαλε. Κάθε κράτο Μέλος κινήθηκε αυτόνομα και είπα ότι εκπρόσωπο η Βαρόνι Άστον δεν μπόρεσε να χειριστεί την κρίση. Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειψε την Ιταλία σε μια ανεξέλεγκτη διείσδυση εισβολή των άστων ε, Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Μάρτιν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ανησυχίες των Ευρωπαίων είναι όλο και πιο μεγάλες επικρατεί μεγαλύτερος φόβος. Και υπάρχουν δύο θέματα τα οποία ε, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Καταρχάς, ε, η ευρωπαϊκή κρίση, η χρηματοπιστωτική κρίση και η μη συνεπής αντιμετώπιση της ύστερα το Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι πίσω από τις εξελίξεις. Ας δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε περικοπή του χρέους τουλάχιστον στην Ελλάδα, ίσως και στην Πορτογαλία δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό το θέμα είναι ότι όσο καθυστερούμε τόσο πιο μεγάλο είναι το κόστος και οικονομικά αλλά και σε ό,τι αφορά την καταράκωση της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό οικοδόμητο. Αυτό που εξακολουθεί να συμβαίνει στην Ελλάδα είναι και πήγαμε και το είδαμε επί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ότι ευθύνεται για τα χρέη στην Ελλάδα γιατί δεν είναι σαφής η επικοινωνία σε ό,τι αφορά τα προβλήματα. Το δεύτερο θέμα, σε ό,τι αφορά την ατομική ενέργεια, τα stress test έχουν νόημα και θα προκαλέσουν και αξιοπιστία, αν θέλετε, μόνο αν αυτές οι δοκιμές αντοχής όντως πληρούν αυστηρά κριτήρια και όχι τα ήπια κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν συμμετέχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και αν τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας δημοσιευτούν με τρόπο κατανοητό. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μάουρο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Στο όραμά μου για την πολιτική πρέπει να προσπαθήσουμε να συναθρήσουμε τα ιδεώδη με τα συμφέροντα. Είναι ένα όραμα ίσως κάπως σχηματικό, αν θέλετε, ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Να τα παρουσιάσουμε σκητσογραφικά. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργάνα εκπροσωπεύουν τα ιδεώδη μας και οι κυβερνήσεις μας για πολλούς λόγους εκπροσωπούν τα συμφέροντά μας. Υπάρχει ένα παιχνίδι που θέλουμε να παίξουμε εδώ. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι θεωρώ ότι σε κάποιες περιστάσεις οι παίκτες ε, του παιχνιδιού των ιδεωδών αρνούνται να παίξουν το παιχνίδι, να κατέβουν στο Εδώ και μερικές εβδομάδες η κυρία Άστον εδώ όταν το Κοινοβούλιο έκανε την πρόταση αναγνώριση ή καλύτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στο Συμβούλιο να αναγνωριστεί το προσωρινό Συμβούλιο της Λιβύης είπε ότι αυτό δεν ήταν η δική της εντολή. Χτες μετά από μια ωραιότατη ομιλία η Επίτροπος Μάλστρομ όταν έφτασε στο ψητό να κάνει πρόταση δηλαδή στο Συμβούλιο μια στρατηγική που θα κάνει η Ευρωπαϊκή την κρίση των μεταναστευτικών ροών είπε ότι παρετείται από αυτό διότι θεωρείται στο Συμβούλιο δεν υπάρχει τέτοια πλειοψηφία. Όμως η ομάδα των ιδεωδών πώς καταφέρνει να νικήσει το μάτσο αν οι παίκτες μας δεν θέλουν να σουτάρουν προς το τέρμα διότι πιστεύουν ότι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα βασικό θέμα για να καταλάβει κανείς ιστορικό πώς τις, ε, το τι καλούμε θα να κάνουμε. Επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την παρατήρηση λοιπόν. Ποιοι είναι οι παίκτες, οι επιθετικοί, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρόεδρος εσείς κύριε Βαν Ρομπόη. Διότι νομίζω ότι εκπροσωπείτε το Συμβούλιο με την έννοια ότι υποσπίζετε τα συμφέροντα. είστε κάποιο που μπορείτε να κάνετε στο Συμβούλιο να καταλάβει ποια ιδεώδη πρέπει να επιδιώκει. Σα ρωτώ απλά λοιπόν, είσαστε παίκτε επιθετικοί μα. Δώστε την μπάλα, περάστε μια πάσα. Παίξτε επίθεση. Βάλτε κανένα γκολ, όπω λέμε σε αυτού του είδου. Κάντε μα να ονειρευτούμε τέλο πάντων. Ευχαριστώ κύριο Γκουαλτιέρη για δύο λεπτά. Αναμφισβήτητα τα, αυτός ο μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας υποστήριξης είναι σημαντικό αποτέλεσμα που δίνει μια βάση στην πολιτική δέσμευση να υπερασπιστούμε πάση θυσία το κοινό νόμισμα. Και γι' αυτό παρά κάποιε επιφυλάξει από τη μέθοδο και την κυβερνητική φύση του Ταμείου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτή την λύση και επικεντρώθηκε από το στόχο να εγγυηθούμε στενή διασύνδεση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Νομίσματος και του Ευρωπαϊκού, ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλαμε ένα κανονισμό για να καθορίζονται οι διαδικασίες που θα καθορίζουν την αιρεσιμότητα και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επεξεργαστεί μια πρόταση ανάλογη που θα υποβάλει. Όμως είναι δύσκολο να δούμε αυτό το αποτέλεσμα σαν θετικό και επαρκές. Ε, το πρόβλημα είναι ε, η κατεύθυνση ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Τι κατεύθυνση. Προσπαθεί να θεραπεύσει τα συμπτώματα της ασθένειας και όχι τα αίτια. Τα ελλείμματα είναι το αποτέλεσμα και όχι το αίτιο της κρίσης και το να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε την ασθένεια περιοριζόμενη στην περιμείωση με το ένα χέρι των ελλείμματο και χρηματοδότηση τραπεζών από την άλλη, είναι αυταπάτη. Υπάρχει κίνδυνο επιδείνωση τη κρίση και να γίνει μη βιώσιμη μη βιώσιμο ο ίδιο μηχανισμό τη στήριξη, ο μόνιμο μηχανισμό στήριξη. Αν θέλουμε λοιπόν να θεραπεύσουμε την ασθένεια και όχι μόνο τα συμπτώματα, θα πρέπει να κόψουμε κάποιου γόρδιου δεσμού. Μιλάμε για ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα Ευρώπη, σωστό, αλλά ποιο μοντέλο ανταγωνιστικότητα επιδιώκουμε. Ε, δεν μπορούμε να ακολουθούμε το μοντέλο μια ανάκαμψη που θα εξαρτάται μόνο από τις εξαγωγές προς το εξωτερικό της Ευρώπης, διότι κάτι τέτοιο θα τονίσει τις ανισορροπίες και για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί ένταντι του εξωτερικού θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε ζήτηση εσωτερική για την ποιότητα. Λοιπόν, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το χρήσιμα τη πίστος, τη δανειοδότησης από πλευράς των τραπεζών, ούτω ώστε οι ευρωπαϊκές οικονομίες να πάνε προς χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Χρειάζεται ευρωομόλογα, χρειάζεται ε, φορολόγηση των χρηματοστικών συναλλαγών για να χρηματοδοτήσουμε ε, ευρωπαϊκά σχέδια, όχι μόνο το ιδιωτικό τομέα. Και χρειάζεται ευρωπαϊκό κοινωνικό, ε, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να μην θεωρείται βάρος, αλλά σαν πηγή. Ο κύριο Μπόλ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Η ε, κυρία Μπολ, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το σύμφωνο Eurosyn μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελέσει ε, ε, δικαιολογία για την ε, αδυναμία του προηγούμενου πακέτου. Η ισχυρή δέσμευση στην ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωζώνη. Αλλά οι πρωτοβουλίε τη ενιαία αγορά παραμένουν στο πλαίσιο τη συνθήκη και των 27 κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αυτό ο μηχανισμό στήριξη νομίζω ότι δεν έχει την επαρκή ευελιξία και ούτε είναι βιώσιμο για την ανάκαμψη με αυτό το ε, κινδύνου του 2,5-3%. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρξει πειθαρχία, αλλά αυτοί οι μηχανισμοί διάσωσης ε, δεν έχουν στόχο την ε, ε, επίτευξη κέρδους οικονομικού, αλλά την σταθερότητα της Ευρωζώνης. Έχουμε σήμερα η στήριξη πολλών τραπεζών από τους φορολογούμενους, παραδείγματος χάρη όπως αναφέρθηκε. Δεν έχουμε λύσει την τραπεζική κρίση, ούτε θα τη λύσουμε εάν δεν αναλαμβάνουμε τολμηρά μέτρα. Ούτε η Γερμανία έχει οδηγήσει στην επανακεφαλοποίηση των τραπεζών τη, ούτε έχει αναγνωρίσει κάποια ε, τοξικά προϊόντα. Και επίση ε, δεν χρειαζόμαστε αντιμετώπιση ανεπαρκή. Πρέπει, αλλιώς θα αποτύχουν οι δοκιμές αντοχές. Επίσης θα πρέπει να είμαστε κάπως ταπεινόφρονες όταν κάνουμε κάποιες κριτικές Νομίζω ότι θα πρέπει αυτά τα ασφάλιστρα κινδύνου να αντιμετωπίσετε ω εγγυήσει. Δεν θα πρέπει να είμαστε κοντόθωροι, δεν θα σώσουμε ούτε το ευρώ και με αυτόν τον τρόπο και το γνωρίζουν και οι αγορέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σέφνερ, έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι καθήκον της πολιτικής ε, με λεφτά των φορολογουμένων να διασώζει τράπεζες και να δημιουργεί ρευτότητα είναι καθήκον της πολιτικής να δημιουργεί τους κατάλληλους όρους πλαίσιους προκειμένου να μην παρουσιαστεί μια τέτοια κατάσταση. Και τώρα καλείστε να κάνετε το εσφαλμένο επειδή επί δεκαετίες δεν κάνατε το σωστό. Και τώρα αυτό που θέλετε, το καλωσορίζουμε αυτό, είναι να αντιμετωπίζετε τα αίτια. Αλλά από ό,τι φαίνεται το κάνετε στο λάθος επίπεδο, με τα λάθος μέσα και στο λάθος πλαίσιο αυτό. Γιατί θέλετε να το κάνετε εκτός των συνθήκων. Ευτυχώς υπάρχει ε, ένα ε, σημείο. Στην κλασική πολιτική θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση, έλεγχος και συζήτηση καταρχάς. Το κάνετε όμως αυτό με τα λάθος μέσα, γιατί παίρνετε τα χρήματα του φορολογούμενου για να διασώσετε και να υποστηρίξετε τις τράπεζες και όσους ε, κερδοσκοπούν μέσω των τραπεζών, αλλά δεν έχετε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να στοχεύσετε αυτούς που έχουν πετύχει κέρδη επί μακρόν. Και έτσι δημιουργείται μια εσφαλμένη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδυναμώνει την πολιτική του μέλλοντος. Αφήνεται τα δημόσια ταμεία, ε, μάλλον ε, επιτίθεται τα δημόσια ταμεία και αφήνεται ε, ελεύθερου του ιδιώτες. Και έτσι αντιμετωπίζεται μόνο τα συμπτώματα, όχι τα αίτια. Ευχαριστώ ο κύριος Φαντάλαν για ένα λεπτό επί σειρά ετών κράτη-μέλη ε, ασκούσαν πολιτική τα οποία, η οποία ε, έκαναν τα δημόσια χρέη να εκτοξευθούν στα ύψη. Το ίδιο έκαναν και οι δυο ε, αγόραζαν ακριβά σπίτια πολύ πάνω από τον προπολογισμό τους. Και πλέον αυτό, αυτή η φούσκα έχει σκάσει. Η κρίση αυτή η φυστάμενη αντιμετωπίζεται με νέα χρέη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγόρασε σε Πορτογαλία, Ελλάδα και η Ιρλανδία ομόλογα τεράστιου ύψους. Επί σειρά ετών θα πρέπει να υπάρχει τεράστια ανάπτυξη για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δεν, πρόκειται να γίνει αυτό. Συρρυκνώνονται οι οικονομίες. Ε, προς πτώχευση οδεύουμε. Έχει λοιπόν έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε την ε, κατάσταση. Θα πρέπει οι χώρες να επανέλθουν, οι χώρες επιτοχευμένες να επανέλθουν στο νόμισμά τους και να δούμε τι θα συμβεί. Ευχαριστώ κυρία Φιγκρέιδο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά και μας φοβίζει αλλά είναι και αποκαλυπτικό αυτό που βλέπουμε ότι οι εκπρόσωποι, οι βασικοί του Συμβουλίου και της Κομισιόν φαίνεται να αγνοούν τη σοβαρή κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζουν ε, χώρες της Ευρωζώνης κυρίως. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους ε, που υποφέρουν από τη φτώχεια. Τι κάνουμε για αυτούς. Πάνω από 20 εκατομμύρια από αυτούς ε, ζουν με πολύ χαμηλούς μισθούς, εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Από την άλλη βλέπουμε τα τεράστια κέρδη των χρηματοοικονομικών ομίλων τι θα κάνουμε για τους ε, νέους ανέργους, τα εκατομμύρια επίσης ε, γυναικών που δεν έχουν μπροστά τους ε, ένα αξιοπρεπές μέλλον, που δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των χωρών τους γιατί δεν έχουν δουλειά. Τι κάνει το Συμβούλιο. Μόνο προασπίζει τα συμφέροντα μεγάλων ομήλων, συγκεντρώνει περισσότερο την εξουσία συγκεντρώνει την οικονομική ισχύ στα χέρια ολιγών και ολιγότερων. Άρα μεγαλύτερη οικονομική κρίση, μεγαλύτερη εκμετάλλευση, λιγότερα δικαιώματα και χώρες όπως η Πορτογαλία να υποφέρουν περισσότερο. Το κύριο ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, θεωρεί το Συμβούλιο Κεντρική Ρύθμιση των Εθνικών Δημοσιονομικών σαν κάτι πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάκαμψη και πιο συγκεκριμένα η πρόταση για πολιτικό σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης που καλύπτει και τα ελλείμματα και έσοδα και έξοδα να πρέπει να υλοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος με κυρώσεις αν δεν γίνει αυτό. Το έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διευθυντικό και θα πρέπει εσωτερικά να λυθεί. Είμαι αντίθετο σε ανάμειξη των Βρυξελών στι υποθέσει τη χώρα μου. Λαμβάνοντα υπόψη τα χάλια που έκανε και στην Ελλάδα στην Ιρλανδία και την ανάγκη για περισσότερε ενισχύσει. Η Πορτογαλία καλύτερα θα στρέφεται προ την Βραζιλία, διότι η Λισαβόνα δεν θέλει να γίνει οικονομικό προτεκτοράτο με, οικονομικ... με μέτρα λιτότητα που θα πνίξουν την ανάπτυξη. Θα πρέπει λέει, να, να δημιουργηθούν μεγάλα ελλείμματα για να προχρηματοδοτηθεί η οικονομική εξυγίανση στα κάτι μελη και θα φύγουν τελικά οι διάφοροι λέει, θα μεταναστεύσουν προ τι ισχυρότερε οικονομίε Ευρώπη. Λέει ότι το διοικητικό άκτο θα πρέπει να μειωθεί, λέει το Συμβούλιο. Μέσω τη νομοθεσία την οποία εθέσπισε όπω το ράδιο εργασία και για την ε, άδεια μητρότητα. Χρειάζεται να είναι πιο ελεύθερα τα μέτρα που υπάρχουν για να μπορεί να κινηθεί η αγορά και όχι να πνίγονται από τα μέτρα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κύριο Μέλτσορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευρωπαϊκή Σύνοδος του Συμβουλίου συζήτησε τρία θέματα αλλά χαρακτηρίζεται από απώλεια της αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά ε, το ένα, τα 100 εκατομμύρια σε ό,τι αφορά το, ταμείο, το, το, το μηχανισμό σταθεροποίησης. Θεωρώ ότι δεν είναι αποτελεσματική αυτή η αντιμετώπιση και έχει πολλαπλασιαστεί ο κίνδυνος αποτυχίας. Κατά δεύτερον, ε, αμφισβητούμε κατά πόσο η αντιπολίτευση του Καντάφη πραγματικά θέλει δημοκρατία. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η στάση του ε, επικεφαλής των ε, ε, δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Τέλος, χάνεται η αξιοπιστία προς τις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά και την ε, εκ νέου δραστηριοποίηση, εκ νέου εφαρμογή μιας ε, νομοθεσίας 20 ετούς σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Δύο λεπτά, κύριε Λαμασούρ. Ένα ή δύο. Δύο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, ε, κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την ΟΚΙ, το αποτέλεσμα του Συμβουλίου είναι εντυπωσιακό. Συγχαρητήρια. Αλλά Λαμβάνοντα υπόψη ότι δημιουργούνται νέα και πολύ σοβαρά προβλήματα, η πολιτική αποδοχή ε, των αποφάσεων πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα. Πρώτον, μεταξύ των ίδιων των κρατών μελών. Ευθύς εξ αρχής η διαδικασία αυτή του ε, συμφώνου Europlus βασίζεται σε μια ε, κυβερνητική ε, αποδοχή με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους. Πάει καλά για μια φορά, αλλά αν επί πολλά χρόνια έχουμε την ίδια πολιτική πορεία θα οδηγηθούμε μάλλον σε σημαντικές εθνικές εντάσεις. Ήδη η Γερμανίδα καγκελάριος ε, γιουχαρίστηκε και στους δρόμους του Δουβλίνου και ε, σε άλλε πρωτεύουσε. Θέλουμε λοιπόν μια αυθεντική ευρωπαϊκή διαδικασία, όχι που δεν είναι ακόμα κοινοτική, αλλά ευρωπαϊκή. Και γι' αυτό ενέκρινε κάποιε σχετικέ τροποβουλίες στο Κοινοβούλιο. Ο Γιούγκερ και εσεί, κύριε Φοντρομπάη πρέπει, επειδή τι εγκρίνατε, να σα συγχαρούμε. Τώρα, δεύτερο επίπεδο. Αποδοχή από την κοινή γνώμη σε κάθε ένα από τα κράτη-μέλη. Πώς τα κόμματα της αντιπολίτευση στις χώρες μας θα ε, ταυτιστούν με αυτούς τους πολιτικούς προσανατολισμούς για τους οποίους όμως δεν στήθηκε ποτέ η γνώμη τους. Ας δούμε τι έγινε χθε ε, στις Ιρλανδικές εκλογές. Ας δούμε σήμερα την ε, συζήτηση που γίνεται στο πλαίσιο των μελλοντικών εκλογών στην Πορτογαλία. Θα πρέπει να δώσουμε στις συστάσεις αυτές ένα είδος πολιτικής νομιμότητας και θα πρέπει εθνικά κοινοβούλια επίσης να συμμετέχουν από την πρώτη μέρα και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όμω αναφέρουν μόνο εν παρόδο τα κοινοβούλια και τα βάζουν στην ίδια κατηγορία με κοινωνικούς εταίρους, περιφέρειες, ΜΚΟ αλλά διακυβεύονται πολύ σημαντικότερα πράγματα. Μιλάμε για μια νέα διάσταση τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Αυτή την οδό πρέπει να διερευνήσουμε. Αυτό μα καλούν να κάνουμε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ δύο λεπτά κύριε Μπούλμαν. Κυρία Πρόεδρε, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μας προτείνουν να ενισχυθούν τα δημοσιονομικά στην Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Αυτό που λέμε εμείς ε, επί του παρόντος, κοιτώντας τι γίνεται και πώς θα λειτουργήσει το, στο μέλλον αυτό, γίνονται λάθος ε, ε, κινήσεις, απολύονται οι επιστήμονε για περικοπέ στον δημόσιο προπολογισμό. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Μπαρόσο, τον κύριο Φανρόμπα, αυτό εννοείται. Θα μου πείτε βέβαια ότι όχι, δεν εννοείται αυτό, ότι κάτι άλλο θα πρέπει να περικοπεί. Ε, μα πού να περικοπεί σας ερωτώ. Και το βασικό μου ερώτημα είναι το εξή. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να γίνουν περικοπές κάπου αλλού, γιατί τα κείμενα τα οποία ε, μας παρουσιάζονται για το πακέτο και την οικονομική διακυβέρνηση δεν είναι σε θέση να κάνουν μια διάκριση κατά πόσο μια χώρα αγοράζει τάγκ, αγοράζει ε, όπλα και επενδύει σε μια λυπηρή κατάσταση ή κατά πόσο επενδύει σε ένα μελλοντικό ενεργειακό σύστημα, κατά πόσο επενδύει στην επένδυση και την κατάρτιση των παιδιών των. Αυτά τα κείμενα είναι χαζά, είχε πει κάποτε ο πρώτη και είχε δίκιο, γιατί δεν μπορούν να κάνουν μια τέτοια διάκριση. Έμα ε, να τα βελτιώσουμε τα κείμενα αυτά. Ιδάλω, δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε σωστά την Ευρώπη, αν δεν μπορούμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Και τελευταία ερώτηση, από πού θα έρθουν τα έσοδα προκειμένου να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε από κοινού και να ξεπεράσουμε την κρίση. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομίες για να ξεπεράσουμε την κρίση. Και περιμένουμε λοιπόν κύριε Μπαρόσο την πρότασή σας για τον Ευρωπαϊκό Φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όπως υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Ας δώσουμε λοιπόν μια καλή ευκαιρία στην Ευρώπη Ευχαριστώ και το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κλίντς για ένα μισή λεπτό. κύριοι πρόεδροι. ακούγοντας προσεκτικά αυτά που λέτε, φαίνεται ότι τα πάμε καλά και ότι το ευρώ έχει διασωθεί και ότι έχουμε ένα νέο πακέτο σταθερότητας και όλα καλά, όλα ωραία. Να σας πω ότι δεν το πιστεύω αυτό. Να μην ξεχνάμε το σημείο εκκίνησης για την όλη κατάσταση, το μεγάλο χρέος μερικών κρατών μελών την χαμηλή ανταγωνιστικότητα και το ότι το νέο πακέτο σταθερότητας δεν μπορούν, ε, προβλέπει όρους που δεν μπορούν να πληρωθούν όσο και να θέλουν κάποια κράτη-μέλη. Κανείς δεν θέλει να χρεοκοπήσει ένα μέλος της Ευρωζώνης και επειδή η προοπτική για χρηματοπιστωτική βοήθεια είναι δύσκολη. Άρα, de facto, είναι εύκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Ξέρουμε ότι το σύμφωνο για το ευρώ είναι πολύ μη δεσμευτικό προκειμένου να περάσουν οι αλλαγές που χρειάζονται Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι δεν θα ε, καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε. Θα υπάρχει μια διευκόλυνση ε, των πιστώσεων διαρκής, ένα πηγάδι χωρίς ε, πάτο και οι πολίτες όλο και πιο πολύ απογοητεύονται και όλο και πιο πολύ μειώνεται η εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έπινγκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία προσωπική ερώτηση έχω να κάνω για τον κύριο Φαρόμπαϊ. Ο πόλεμος στη Λιβύη συνεχίζεται. Είδαμε τις στενές σχέσεις μεταξύ του ηγέτη της Λιβύης και ε, των ε, Ευρωπαϊκών Προέδρων. Σας εκτιμώ κύριε Φαρόμπαϊ. Είσαστε άνθρωπος ακέραιος ακόμα και στην πολιτική. Είσαστε συνεπεί. Γι' αυτό με ενόχλησε λοιπόν πάρα πολύ αυτέ οι φωτογραφίε δολοφονείται κόσμος με όπλα ευρωπαϊκά και βλέπουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες με τον ε, δολοφόνο. Με απογοητεύσατε λοιπόν. Ίσως επειδή είστε καινούριο στη θέση αυτή, αλλά θα ήθελα να σας συστήσω να είσαστε πιο σταθερός στην πολιτική σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιλέξει την πλευρά της ελευθερίας. Και αυτό διακυβεύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και ο κύριος Μπαρόσο επίσης, επίσης ήταν πάρα πολύ ε, φιλικός προς τον δικτάτορα. Με απογοήτευσε επίσης. Ευχαριστώ ο κύριος Φεκμαρ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μέχρι τώρα είχαμε αντιμετωπίσουμε την κρίση με το χρέος Και τώρα πρέπει να ασχοληθούμε τα αίτια, τα θεμελιώδη προβλήματα που δημιούργησαν ε, την κρίση, τα τεράστια λύματα και τα αδύναμα δημοσιονομικά. Και γι' αυτό ε, αυτό το σύμφωνο σταθερότητας είναι υψής της σημασίας. Όχι μόνο για να πετύχουμε τους στόχους, αλλά για να δημιουργηθεί και κάποια αξιοπιστία για τις οικονομίες της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε επίσης αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων, δηλαδή έλλειψη ανταγωνιστικότητας, έλλειψη οικονομικής αναπτύξεως. Αυτό είναι το βασικό μας έργο για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να δημιουργήσουμε απασχόληση και να εξασφαλίσουμε την ευμάρεια. Τα κράτη-μέλη υπέχουν ευθύνες εδώ. Πρέπει να αναδιαστρώσουν τους προϋπολογισμούς και να δώσουν προτεραιότητα στην κοινωνική ασφάλεια και επενδύσεις ταυτόχρονα για την ανάπτυξη, όσο μειώνονται τα έλλειμματα. Χρειάζεται επίσης μεταρρύθμιση των αγορών, αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν και δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη και πολλά περισσότερα. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε επίση το τι θα πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είμαστε εξίσου έτοιμοι να αναδιαθρώσουμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, κάτι που απαιτούμε από τα κράτη-μέλη. Να εξασφαλίσουμε ότι θα δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη, στι επενδύσει, στην έρευνα, στι επιστήμε και στι ανοιχτέ αγορέ και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση το ότι μεταρρυθμίζουμε τι ευρωπαϊκέ αγορέ. 70% τη ευρωπαϊκή οικονομία είναι ο τομέα των υπηρεσιών. Η οδηγία των υπηρεσιών είναι αρκετά περιορισμένη όσον αφορά αυτή την προοπτική. Το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας έγκυται στον τομέα της, ε, των υπηρεσιών και στον τομέα της οικονομίας της γνώσης. Και υπάρχει έτοιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που θα καθιστούν την, Ευρωπα... την ενιαία αγορά εφαρμόσιμη σε όλο τον τομέα των γνώσεων. Θα πρέπει να γίνει η ηγούμενη στον κόσμο οικονομία της γνώσης η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπερές έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μετά την κρίση αυτή για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, ποιο είναι το όπλο το καλύτερο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο σας το είπατε, η στρατηγική για την Ένωση, η στρατηγική 2020. Βλέποντα αυτά που κάνετε στα θέματα τη οικονομική διακυβέρνηση, βλέπω πάντω να υπάρχει απόλυτη αντίφαση. Διότι α δούμε το Σύμφωνο Σταθερότητα, οικονομική διακυβέρνηση. Από μια στρατηγική συντονισμού τίνεται να περάσετε σε μια στρατηγική εποπτείας, επιτήρηση η οποία μεταφράζεται στην, ε, σε έναν, από συνένεση της Ουάσιγκτον σε συνένεση των Βρυξελών. Όταν μιλάτε για διαφορετικέ μεταρρυθμίσει. Μιλάτε για μείωση των μισθών, αύξηση του ορίου συνταξιοδότηση. Εγώ θα σα μιλήσω όμω για τι πραγματικέ διαφορετικέ μεταρρυθμίσει που χρειαζόμαστε. Δημόσιε επενδύσει πρώτα απ' όλα. Πρώτον στην εκπαίδευση. Ξέρετε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτή τη στρατηγική τη Λισαβόνα το ίμιση των κρατών μελών μείωσαν του προπολογισμού του ε, για την παιδεία. Επιβάλλατε καιρό σε αυτά τα κρατημέλη. Για αυτό το λόγο. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν θα υλοποιεί στρατηγική 2020 εάν δεν έχουμε κάποιες κοινέ επενδύσεις για το μέλλον, εάν εξαιολογείς τις δημόσιες δαπάνες των κρατών, θα δείτε ότι στις μόνες δαπάνες που κάπως υπάρχει διαφορετικό μάτι, ε, που βάζετε ποιοτικό στοιχείο εκεί, είναι η ε, μεταρρυθμίσεις ε, των συντάξεων με της κεφαλαιοποίησης. Λέτε ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες. Τι θα κάνουμε στον τομέα της παιδείας, αν δούμε την κατάσταση σήμερα στην Ιρλανδία. Εμένα εκεί με εκπλήσει το εξή και με εντυπωσιάζει ότι κάθε μέρα αποφασίζουμε να διασώσουμε κάποια τράπεζα. Οι Ιρλανδοί όμως τελικά μας εγκαταλείπουν λίγο-λίγο. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε. Εγώ νομίζω ότι καλύτερο είναι να σώσουμε τον Ιρλανδό παρά την τράπεζά του. Και για να σώσουμε τις τράπεζες έχουμε επινοήσει τον όρο stress test, αυτές τις δοκιμές αντοχής. Και έχω την ότι κάθε φορά που προκύπτει δυσκολία πετάμε και ένα stress test. Είναι ε, η νέα ε, επιτροπή stress test για τις τράπεζες, stress test για τα πυρηνικά, stress test και για την Κομισιόν αύριο. Ναι, πράγματι, γιατί όχι, ίσως να το προτείνουμε και αυτό. Αλλά εγώ αυτό που θα προτιμούσα θα ήταν μια Κομισιόν που θα παίρνει πρωτοβουλίες και που θα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Βλέποντα τι γνωμοδοτήσει τη της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα, βλέπω να ανησυχεί για κάτι που δεν είναι στην εντολή τη, δηλαδή για του μισθέ και όχι για την βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματο και για τι δημόσιε επενδύσει που χρειαζόμαστε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει κάποιε προτάσει. Αρνείστε να τι λάβετε υπόψη φορολογία χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ευρωομόλογα. Κύριε Πρόεδρε, είναι καιρό να ακούσετε τι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υλοποιήσετε και την ίδια στρατηγική που προτείνετε. Διακόπτη πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Εκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Ο Πρόεδρος ε, μίλησε και την προηγούμενη φορά για το θέμα της ασφάλειας των ε, πρινικών σταθμών και των πρινικών αντιδραστήρων. Πρόκειται ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης στο Κοινοβούλιο. Θα υπάρξει ένα ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί τελικά την Πέμπτη. Ως Ευρωπαία πολίτης θεωρώ ότι πολλοί θα θεωρούσαν ότι ασφαλώς και υπάρχουν δοκιμές αντοχές ως τμήμα, αντοχής, ως της πολιτικής για, τα πρινικά, για τους πρινικούς σταθμούς, το οποίο δεν ισχύει όμως και αναφέρεται πάρα πολύ αδύναμα λόγια στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα πρέπει να ελέγξουμε και την όλη κουλτούρα της πολιτικής ασφάλειας. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει διαφάνεια και είναι απόλυτα αδυνατό σε αυτό το πλαίσιο οι εθνικές αρχές να ελέγχουν τα στοιχεία αυτά. Αυτό θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονε. Όλα θα πρέπει να δημοσιεύονται με πλήρη διαφάνεια, με δυνατότητα ελέγχου της Επιτροπής. Η μοναδική ευκαιρία είναι αυτή για να διαμορφώσουμε με αξιόπιστο τρόπο την τεχνολογία αυτή. Χρειαζόμαστε ε, μία ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα είναι τόσο παλιό όσο και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, θα πρέπει να φροντίσουμε και το Υπουργικό Σύμβουλιο να υποβάλει τέτοιε προτάσεις σε ό,τι αφορά τη ενεργειακή αποδοτικότητα και τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Και διακόπτει η Πρόεδρος. Ναι, 1,5 λεπτό είχατε το λόγο, όχι 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. κυρία Φόρτ. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα του Συμβουλίου δεν ήταν σε έξι για του τίτλου των εφημερίδων. Είπε ότι η νέα αγορά έχει βασικό ρόλο διαδραματίσει για να πετύχει την ανάπτυξη. Αλλά είναι όλα αυτά λόγια. Όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, ήδη βλέπω ότι κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να αποδυναμώσουν το σύμφωνο σταθερότητα. Και όσον αφορά την υποστήριξη των επιχειρήσεων, δεν τα κάνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Οι ευρωβουλευτέ θέλουν να υπογράψουν εκστατείε υπέρ των ποδηλατών ε, και άλλου για άλλου στόχου. Όταν όμω θέλανε για περικοπή ε, τη γραφειοκρατία μικρομεσή μόνο το 1 τρίτο συμμετέχει και μόνο μη υπογραφή από το Εργατικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασίλειου Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως ε, θέλει να απελευθερώσει τις επενδύσεις κεφαλαίου. Αξιέπαινο, αλλά άμα δείτε τι ξοδεύτηκε πέσει για να νομοθετηθεί εκτός αγοράς αυτό το κεφάλαιο είναι γελίο σήμερα. Οπότε πρέπει να γίνουν πράξη αυτά που λέγονται. Νέα αρχηγοί κατών κυβερνήσεων υπέγραψαν επιστολή με συγκεκριμένε δράσει για την εμπόριο, την καινοτομία, τι επενδύσει και τι επιχειρήσει. Μα ζητούν επιλέξουμε την ανάπτυξη και εγώ σίγουρα το επιλέγω. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μία δέσμη μέτρων σε σχέση με την ε, διακυβέρνηση, τη δημοσιονομική εξυγίανση, την ανταγωνιστικότητα και θέλω να πω ότι όλα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτά τα 16 σημεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε μεγάλο βαθμό οφείλονται, χάρη, ε, οφείλονται σε αυτό που έκανε και ο πρόεδρος Φοντρόμπα και ο πρόεδρος Μπαρόσο στις προσπάθειές τους και γι' αυτό πρώτον πρέπει να τους συγχαρώ γιατί εγώ κάποιοι από εμάς εκτιμούμε αυτά που είπατε. Όμως κύριε πρόεδρε δεν πρέπει να ξεχνάμε πρόκειται για μια οικονομική κρίση αλλά και για μια κρίση εμπιστοσύνης, μια κρίση που έχει πολιτικό χαρακτήρα για την Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχέσεις. Και δεν μιλάμε μόνο για συγκεκριμένες οικονομικές και τεχνικές αξίες και όρους. Υπάρχουν ε, και εθνικές ε, και περιφερειακές ευρωπαϊκές εκλογές. Και σε όλες αυτές βλέπουμε ότι υπάρχει ε, εκνευρισμός. Υπάρχουν ακραίες θέσεις. Υπάρχουν μέχρι και εθνικιστικές τάσεις σήμερα. Και νομίζω ότι εσείς πρέπει να καταλάβετε σήμερα ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε όχι μόνο την κρίση αλλά και τις πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Δεν έχουμε μόνο μια κρίση βορρά-νότου, όπω πολύ σωστά είπε κάποιο ε, συνάδελφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι νέοι καιροί. Είναι μια νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από τη συσσόρευση και τον πολλαπλασιασμό των κρίσεων που δεν επιλύονται και αναδύονται έτσι έφνης και εντός και εκτός. Απαιτείται λοιπόν νέα, νέα συμπεριφορά, νέα... Ε, νέοι θεσμοί. Και αυτή είναι η πολιτική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε τις νοοτροπίες και τη θεώρησή μας και εμείς και θα πρέπει να πούμε πώς πρέπει να αλλάξουμε για να αντιμετωπίσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτούς τους νέους καιρούς. Και το ίδιο πρέπει να το κάνει και η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όλοι πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα κατάσταση. Πάντως ε, πρέπει να ξέρετε ότι πάτε προς σωστή κατεύθυνση, συνεχίστε έτσι. Ο κύριος Σάντσες, πρεσέντο για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόκειται για την πρώτη κρίση της Ευρωζώνης. Ε, όταν ήρθε αυτή η κρίση, είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν κατάληξη όπω σημαίνει για την αντιμετωπίση. Υπήρξαν σφάλματα σχεδιασμού, παραλίγματος ε, χάρη κάποια ε, ε, σε λήψη χρηματοπιστωτικό σύστημα, μη εκπλήρωση δεσμεύσεων στα δημόσια οικονομικά, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, μεγαλύτερε μακροοικονομικέ ανισορροπίε και αποκλήσει εντό Ευρωζώνη. Είδαμε επίση πώ τα βήματα τα οποία είχαν δοθεί για να έχουμε μια ευρωπαϊκή φωνή στο πλαίσιο τη ε, ΚΕΠΑ δεν συνοδεύτηκε με αντίστοιχα πράγματα στον οικονομικό τομέα. Δεν μπορέσαμε εν ώψη της παγκοσμιοποίησης την οικονομική ηγεσία μας να την ε, προωθήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είδαμε πάρα πολλά προβλήματα να ε, προκύπτουν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Δεν υπάρχει εθνική διέξοδος, εθνική λύση. Νομίζω ότι κάποιοι κάνουν λάθος στον αιώνα που βρισκόμαστε. Στις 24 και 25 Μαρτίου το Συμβούλιο έκανε σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, θεαματικά βήματα θα έλεγα μεταξύ άλλων. Παραδείγματο χάρη, δρομολογήθηκε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εγκρίθηκαν, εγκρίθηκε ο μόνος μηχανισμός στήριξης με τι ε, δεσμεύσεις που είχαμε προτείνει και στο Κοινοβούλιο, καθώ και το νομοθετικό πακέτο που θα είναι απαραίτητο. Όλα αυτά είναι θετικά. Τώρα, το, το σύμφωνο Europlus ναι μην είναι πρόοδο, αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη, διότι επιμένει η κρίση. Υπάρχουν 23 εκατομμύρια ανέργων, σημαντικά ε, σύννεφα που σκοτεινιάζουν τον ευρωπαϊκό ουρανό. Τριπλή η διάσταση. Έχουμε μια πολιτική λιτότητα που έχει κάποια όρια. Και θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τις επενδύσεις για να επαναπροσανατολίσουμε το οικονομικό μας μοντέλο και να υλοποιήσουμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η πολιτική φορολογικής και χρηματοπιστωτικής βιωσιμότητας απαιτεί ευρωπαϊκό πλαίσιο και σε ό,τι αφορά το εθνικό χρέος και σε ό,τι αφορά την επανακεφαλαιοποίηση. Διακόπτει ο πρόεδρος. Πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, να έχουμε φορολογική πρόοδο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Τρέτσακ για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα όσα συνέβησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 24 και 25 Μαρτίου και τα όσα εγκρίθησαν στη συνέχεια είναι η ιστορία της επιβολής της φορολογικής Ευρώπης από το παράθυρο και η δημιουργία του ευρώ είναι ε, άγνοια ε, της ιστορίας της οικονομίας και μια ιστορία ψευδών για τα οικονομικά και πώς λειτουργεί η οικονομία. Δεν έγιναν σεβαστά τα όσα ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Βλέπουμε ότι διαφέρουν οι εθνικέ οικονομίες. Είναι διαφορετικό ο πληθωρισμό από χώρα σε χώρα και η απασχόληση και το είδο της απασχόλησης. Τι θέλουμε. Νομίζουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα αλλάξει στα πλαίσια του Συμφώνου για το Ευρώ ΣΥΝ. Ούτε σύμφωνο διακόπτη, Πρόεδρος, για δύο λεπτά ο κύριος Άγγελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ και θα ήθελα καταρχήν να σας ε, συγχαρώ για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου 24 και 25 ε, Μαρτίου και κυρίως για το γεγονός πως παγιώθηκαν τα όσα θα γίνουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Μιλάμε λοιπόν για την θεσμοθέτηση του μηχανισμού στήριξης και επίσης για το σύμφωνο Europlus, τα οποία ε, συμφωνήθηκαν ήδη από την 11η Μαρτίου. Για εμάς τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα θετικά για την Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι κρίμα που δεν έκλεισε η διαδικασία στις 24 και 25 Μαρτίου. Πάντως στείλαμε ένα μήνυμα και αν είχαμε δώσει ένα μήνυμα ακόμα πιο στεναρό ως κράτη-μέλη, δηλαδή αν είχαμε φέρει σε τέλος αυτή τη ριζική μεταρρύθμιση, φαντάζομαι πως η θέση μας ήταν πολύ πιο ισχυρή το επόμενο τρίμηνο, τετράμινο. Γιατί βέβαια πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση που αντιμετωπίζουν κάποια κράτη, όπως το δικό μου, η Πορτογαλία. Να σας πω πάντως πως ε, για το δικό μας ε, κόμμα, το οποίο είναι τμήμα του ΕΛΚ, έχουμε αποφασίσει και έχουμε δεσμευθεί πως θα σεβαστούμε όλες, όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Και μάλιστα, τη στιγμή αυτή όπου οι δυσκολίες για την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση Αντίθετα με τα όσα έκανε η σοσιαλιστική κυβέρνηση, εμείς είμαστε απόλυτα διαθέσιμοι για να δώσουμε τις εγγυήσεις στην Ευρώπη που είναι απαραίτητες στα πλαίσια της σημερινής κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν στέλνω αυτό το μήνυμα, πως η εσωτερική πολιτική η η εσωτερική πολιτική που ακολουθούμε, σας το εξασφαλίζω εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου, θα σεβαστεί πλήρως τις δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει. Για, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι συμφωνία. Ε, είναι και επιτυχία ε, της Ουγγρικής κυβέρνησης, συντηρητική επιτυχία. Ενδιαφέρονται μόνο για την ενότητα, ανεξάρτητα με το τίμημα και είναι λυπηρό που δεν συμμετέχουν στο σύμφωνο για το ευρώ τέσσερι χώρε με συντηρητικέ κατά τα άλλα κυβερνήσει. Τι θέλουμε εμεί, τι περιμένουμε από την Ουγγρική Προεδρία. Να τηρεί τι προτάσει της. Μα όποιο δεν συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια θα μείνει πίσω. Θα πρέπει να βασίσουμε όλοι μας τη δουλειά, τη γνώση, στην καινοτομία, αντί να αλλάξουμε τους κανόνες για τη φορολογία. Στην Ευρώπη θα γίνουμε ήπειρος των φτωχών και τώρα έχουμε και φορολογικό ανταγωνισμό. Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι. Το ε, Συμβούλιο δεν συζήτησε ούτε έλυσε τίποτα σχετικά με τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό δεν επηρεάζει τους Ευρωπαίους πολίτες. Εμείς περιμένουμε πολύ περισσότερα από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεγαλύτερη πρόοδο. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω και την άποψή μου για τις ε, εξελίξεις και τα γεγονότα στην Ιαπωνία. 12.000 νεκροί, πολλές χιλιάδες οι αγνοούμενοι και πάρα πολλοί επίσης οι άνεργοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχεια πρεσβεύει την αλληλεγγύη. Πρέπει να βοηθήσει τώρα. Η καταστροφή αυτή, η θεομηνία στην Ιαπωνία οδήγησε σε σοκ και τις αγορές ενέργειας και θα επηρεάσει και την πολιτική και το περιβάλλον για μεγάλο διάστημα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την πυρηνική ασφάλεια με νέες προδιαγραφές με νέα μέτρα να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη με έμφαση στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Ιδού η στόχοι και συμπεριλαμβάνονται και στρατηγική για την Ευρώπη για το 2020. Τώρα εναπόκειται σε Κομισιόν και Συμβούλιο να το προχωρήσει και σας έχουμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρας, λέει Πρόεδρος, τον οποίο και δεν βλέπω στην αίθουσα. Οπότε θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ποδηματά, παρακαλώ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τη σημασία των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η λογική που χαρακτηρίζει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις εδώ και ένα χρόνο είναι πολύ αργά, πολύ λίγο. Και αυτό όχι γιατί δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τα μπρος, αλλά γιατί το μέτρο σύγκριση σήμερα δεν μπορεί να είναι το παρελθόν, το τι κάναμε παλαιότερα για τη σταθερότητα και την ενίσχυση της ευρωζώνης αλλά το πόσο αποτελεσματικοί είμαστε στην αντιμετώπιση της κρίσης και δυστυχώς δεν είμαστε αποτελεσματικοί ούτε απέναντι στις αγορές αρκεί να δείτε πού έφτασε τις τελευταίες ημέρες το κόστος δανεισμού για τις χώρες της περιφέρειας και ειδικά της πορτογαλίας αλλά δεν είμαστε δυστυχώς αποτελεσματικοί και πιστικοί ούτε απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες που θεωρούν ολοένα και περισσότερο και περισσότεροι ότι η ευρώπη δεν είναι μέρος της λύσης αλλά μέρος του προβλήματος το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με δύο πρόσφατα ψηφίσματά του αλλά και εξέχουσες προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα έχουν επισημάνει ότι για να υπάρξει μια αποτελεσματική και συνολική απάντηση στην κρίση χρέους θα πρέπει να εξετάσουμε στα σοβαρά τη λύση ενός συστήματος έκδοσης ευρωομολόγων και η πλειοψηφία του ευρωπαϊκού συμβουλίου απαντά ότι αυτό δεν γίνεται γιατί σε συνθήκες κρίσης θα δημιουργούσε ηθικό κίνδυνο για τις υγιείς δημοσιονομικά χώρες και ενώ όμως επικαλούνται τον ηθικό κίνδυνο για να αντιστρατευτούν το ευρωομόλογο δημιουργούν ηθικό κίνδυνο σε βάρος των χωρών με οικονομικές δυσκολίες βάζοντας επισήμως στο τραπέζι χωρίς κανένα δισταγμό την προοπτική της ελεγχόμενης χρεοκοπίας και της εμπλοκής των ιδιωτών στον επιμερισμό του κόστους και έτσι διαιωνίζουμε την κρίση κρατώντας σε δυσθεώρητα ύψη το κόστος δανεισμού. εάν θέλουμε ειλικρινά συμμετοχή των ιδιωτών και έναν δικαιότερο επιμερισμό του κόστους τότε να εξατέσουμε στα σοβαρά και κατά προτεραιότητα την επιβολή φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ώστε μέρος των εσόδων να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του μόνιμου μηχανισμού. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κοβάτσεφ. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και να σας πω πως η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα αποδεικνύει πως χρειάζεται οραματιστές η Ευρώπη, όχι μόνο πολιτικούς οραματιστές αλλά και πολίτες με όραμα. Είναι λυπηρό αλλά είναι αληθινό. Έχουμε χάσει ε, πολύ χρόνο. Και βέβαια το ενιαίο νόμισμα είναι σίγουρα μια επιτυχημένη προσπάθεια, αλλά είναι σαν ένα όμορφο οικοδόμημα στο οποίο έχει καταρρεύσει η στέγη. Έχουμε γνωρίσει και επιτυχίες και αποτυχίες, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω πως βρέχει στην Ευρώπη. Το σύμφωνο ε, Europlus και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου μας οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση και ο προπολογισμό θα μα βοηθάει καλύτερα να αντιμετωπίζουμε την κρίση και θα γίνεται καλύτερο συντονισμό. Και πρέπει να σα πω πω και χώρε όπω η δική μου, η Βουλγαρία, θα συμμετάσχουν στο σύμφωνο αυτό έτσι ώστε να επηρεάζουν και αυτέ τη διαδικασία λήψη αποφάσεων έτσι ώστε να μην έχουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Είμαι πεπισμένο πω η πολιτική θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κοινοτικά εργαλεία και όχι διακυβερνητικά. Χρειαζόμαστε ίσως μία νέα συνθήκη, αν όχι μία νέα διακυβερνητική διάσκεψη, για να λάβουμε κάποια νέα οικονομικά και πολιτικά μέτρα. Τώρα, για τη Λιβύη και για τη Μεσόγειο, νομίζω πως χρειάζεται να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να βοηθήσουμε την Λιβύη στην πορεία προς τον εκδημοκρατισμό. Και νομίζω θα είναι ένα θετικό μήνυμα για την περιοχή, όπου θα λέμε πως η Ευρώπη στηρίζει τις νόμιμες διεκδικήσεις των πολιτών να κάνουμε κάτι παραπάνω για τους γειτόνους μας. Μήπως θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη δική μας θετική εμπειρία με τις εταιρικέ σχέσεις που είχαμε αποκτήσει στο παρελθόν έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη λεκάνη της Μεσογείου να αναπτυχθεί. Κύριε Βαν Ρόμπα, κύριε Μπαρόσο, η Ευρώπη χρειάζεται να έχει μια λειτουργική ε, δυνατότητα άμεσης και επίγουσας δράσης και αντίδρασης. Ευχαριστώ κύριος Δαρντέν για δύο λεπτά παρακαλώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Βαν Ρομπόη. Είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποια προφανή στοιχεία στα συμπεράσματά σας. Ε, αυστηρή διακυβέρνηση, όλοι συμφωνούμε, αλλά η αυστηρότητα ή η λιτότητα δεν μπορεί να σημαίνει πραγματική λιτότητα και ανάπτυξη μηδέν. Η απαραίτητη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης πρέπει να ε, βελτιωθεί. Βεβαίως, είναι προφανές, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει ε, προς ζημία των κοινωνικών διεκδικήσεων, καθώς επίσης και την μείωση των μισθών. Ε, ε, η Ευρώπη θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη καμπή. Αλλά δεν θα πρέπει να ομφαλοσκοπεί. Δεν θα πρέπει δηλαδή όλοι να δείξουν εσωστρέφεια ε, σε σχέση με τις σχέσεις με τους γειτόνους τους και προσπαθώντας να συμβάλλουν όσο γίνεται λιγότερο προς την Ευρώπη. Η άλλη επιλογή είναι να επιλεγεί η αλληλεγγύη, το μόνο στοιχείο το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό μια ε, ε, ε, μια αποδοχή των ελάχιστων κοινωνικών κεκτημένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλληλεγγύη διασφαλισμένη μεταξύ <clears throat> των γενεών μέσω ενός συστήματος συντάξεων το οποίο θα είναι δίκαιο όπως κατέδειξε πρόσφατα και το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας ε, τις πιέσει των αγορών. Θα πρέπει επίση οι οίκοι αξιολόγηση να μπουν σε μια σειρά. Θα πρέπει να ελέγχονται επίση επίσης να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μαζί με ε, ταυτόχρονη εκβάθους αναδιάρθρωση του συστήματος των ιδίων πόρων. Τα συμπεράσματά σας βασίζονται σε μια ιδεολογία βάσει της οποίας τα ελλείμματα έχουν δημιουργήσει την κρίση, ενώ στην ουσία είναι οι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι μας οδήγησαν στην κρίση αυτή. Ε, με τα συμπεράσματα αυτά του Συμβουλίου δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση, ούτε θα ξαναδώσουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες. Θέλουμε σαφή δημοκρατία και οι προτάσεις του Συμβουλίου δεν λαμβάνουν υπόψη τους την δημοκρατία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα μας απορρίψουν οι πολίτες της Ευρώπης. Η ε, κυρία Τάισεν έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε κύριοι πρόεδρε, ε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να μπορέσει στο μέλλον η Ένωση να είναι μια κοινότητα όπου αξίζει κανείς να ζει και να εργάζεται αξιοπρεπώς. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους τους συναδέλφους που ε, επένεσαν με τη σειρά τους το Συμβούλιο. Ε, θέλω να πω τα εξή όμως. Το πρώτο έχει να κάνει με το μισθολογικό κόστος, το κόστος εργασίας ως ένα παράγον ανταγωνιστικότητας. Κατά τη διάρκεια της κρίσης απευθύνθηκα και στον πρόεδρο του Συμβουλίου και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους επένεσα για τους ε, αυτόματους σταθεροποιητές. Να έχουμε πιο σταθερή οικονομία χωρίς ε, επιλογή κατά καιρού ότι ο καθένας θεωρεί σκόπιμο. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη σταθερότητα της απασχόλησης. Μερικοί όμως τώρα φοβούνται για το σύμφωνο για το Ευρώσυν ότι περιορίζεται πολύ ο χώρος για τους αυτόματους σταθεροποιητές και θέλω να σας ρωτήσω πώς το αξιολογείτε. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να φέρω. Ακούω συνέχεια από τα συνδικάτα να υποστηρίζουν ότι ε, στους μισθούς θέλουν ε, να ε, περιορίσουν ε, την ευελιξία των κρατών μελών και τους κοινωνικούς εταίρους στη δυνατότητα διαμόρφωσης των μισθών. Και μάλιστα γίνεται λόγος και για κατοχήρωση στη συνθήκη. Αυτό είναι κίνδυνος, δεν είναι. Πώς εσείς το αναλύετε κύριε Προεδρεύον και κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αν αυτός ο διπλός φόβος είναι τεκμηριωμένος και βάσιμος, να το εξηγήσουμε και να το διασκεδάσουμε. Και σε ό,τι αφορά την κοινή φορολογική βάση, ε, για τις επιχειρήσεις. Διαβάζω μία και μόνη πρόταση ε, ελάχιστη και χωρίς καμία δέσμευση στο κείμενο των συμπερασμάτων της Αρινής Συνόδου. Πρέπει να σας θυμίσω ότι υπάρχει συνένεση εδώ και καιρό για κοινή φορολογική ε, βάση και δεν ξέρω, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε την ελευσιμένη συνεργασία. Ευχαριστώ. Κύριος Αρσένης, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του στον πρόεδρο του Συμβουλίου και τη Επιτροπή. Η Άννη Ποντιματά με κάλυψε στο θέμα των οικονομικών. Θα αναφερθώ σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, στο ζήτημα τη πυρηνική ενέργεια. Τι μα δίδαξε η Ιαπωνία. Δύο πράγματα. Ένα ότι κανένα δεν μπορεί να είναι ποτέ επαρκώ προετοιμασμένο για φυσικέ καταστροφέ και συνδυασμού του. Το δεύτερο είναι ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ποτέ απολύτω ασφαλή τι κάνουμε εμείς. Κατηγορούμε την Ιαπωνία για αμέλεια. Λέμε ότι δεν ήταν ε, η πυρηνική ενέργεια αλλά η Ιαπωνία που δεν ήταν ασφαλής. Λέμε ότι θα κάνουμε τους δικούς μας ελέγχους, τα, ακριβώς ε, τα δικά μας τεστ στους σταθμούς της πυρηνικής ενέργειας, να δούμε ποια δεν είναι ασφαλή και ποια είναι ασφαλή και μετά να προχωρήσουμε στη συνέχεια τους και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Δεν πήραμε όμως έτσι τα μαθήματα από την Ιαπωνία δεν έχουμε καν την ετοιμότητα της ιαπωνίας απέναντι στις καταστροφές δεν έχουμε καν την πολιτική για την πολιτική προστασία των πολιτών μας απέναντι σε διασυνοριακά προβλήματα όπως ε, ένα πυρηνικό ατύχημα. Πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε σήμερα την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών. Να επενδύσουμε όχι στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, αλλά στην ανάπτυξη της απόδοσης των φωτοβολταϊκών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι επιπτώσει τη πυρηνική ενέργεια είναι διασυνοριακέ και γι' αυτό είναι και ευθύνη τη ευρωπαϊκή ένωση. γι' αυτό κύριε μπαρόζο κύριε Ρομπόη, θα είναι και δικιά σα μεγάλη ευθύνη αν δεν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε ένα νέο ατύχημα. Το λόγο τώρα έχει ο Έχετε το λόγο, κύριε Σάρισβάσκη. Θα ήθελα να ξεκινήσω σχολιάζοντας τρία θέματα. Καταρχήν, πιστεύω πως η Σύνοδος έδωσε πολύ θετικά αποτελέσματα δεδομένη της δυσκολίας κατάστασης, όπως επίσης και του πλησίου μέσα στο οποίο έγινε η συνάντηση. Χαιρετίζω λοιπόν αυτήν την τόσο ευέλικτη και ε, συμπεριεκτική διατύπωση που έχουμε στο σύμφωνο Europlus. Πολύ σωστά μίλησαν και οι συνάδελφοι και τα όσα είπατε και εσείς γιατί δημιουργεί έναν μηχανισμό σταθερότητας με ένα δίχτυ ασφαλείας. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να δούμε πως και το Europe Plus που είναι μια δέσμευση να γίνουν σεβαστοί κάποιοι μακροοικονομικοί και μακροδημοσιονομικοί κανόνες ε, και ε, το μηχανισμό σταθερότητας να εφαρμοστούν αλλά με κάποια ευελιξία έτσι ώστε να μην αποκλείεται κανείς από αυτό το δίχτυο ασφαλείας. Για την πολιτική καλή ε, γειτονιά πρέπει να σας πω πως αυτή τη στιγμή χρειάζεται να την ξανασχεδιάσουμε και βέβαια το κίνητρο γι' αυτό είναι τόσο συμβαίνουν στο Νότο. Θα ήθελα αυτή η πολιτική, η σφαιρική πολιτική να είναι, εάν διαβάσουμε τα κείμενα Άστον και Φίλερ, να είναι πιο ανοιχτά προς τις τοπικές κοινωνίες, πιο γενναιόδωρα προς τις κοινωνίες αυτές και ίσως και πιο απαιτητικά προς τις κυβερνήσεις και τις αρχές. Νομίζω πως θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τα κοντόφθαλμα οικονομικά συμφέροντα και να βασίσουμε την πολιτική αυτή σε μια προσέγγιση που θα έχει ως αρχές τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών. Να έχουμε και μια πολιτική για τις χώρες που βρίσκονται σε, βρίσκονται σε μετάβαση. Όταν θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα νέα υποδείγματα, τα νέα μοντέλα, να τα εξαπλώσουμε και προς την Ανατολή, έτσι ώστε οι κοινωνίες αυτές να βασίζονται περισσότερο στην κοινωνία των πολιτών και λιγότερο στα όσα επιθυμούν οι αρχές. Και η τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με τις σχέσεις Ευρώπης-ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ. Εδώ έχουμε μια νέα εμπειρία, νέο δίδαγμα από τα όσα γίνονται στη Λιβύη και είναι ίσως κάτι το οποίο ακόμα δεν γίνεται πλήρως κατανοητό. Ε, η εμπειρία μας από το Αφγανιστάν ίσως δεν είναι πάντοτε θετική, αλλά η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι σημαντική, ας είναι λοιπόν επιτυχημένη, τούτη τουλάχιστον τη φορά. Το λόγο έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Κάριντς. για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Και όταν μιλώ για το παρελθόν, πρέπει να βρούμε μία λύση ενιαία για την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος απόσβεσης του χρέους με διαρθρωτικά μέτρα. Θα πρέπει οι κοινωνίες να συνεχίσουν να ζουν και δεν μπορούν να τιμωρούνται οι πολίτες των χωρών αυτών για λάθη και αμαρτίες του ιδιωτικού τομέα και προκειμένου των τραπεζών. Για το μέλλον όμως τώρα θα πρέπει να κοιτάξουμε τι στόχο έχουμε στην Ευρώπη, τι σκοπό έχουμε, να εξασφαλίσουμε σταθερή ανάπτυξη. Πώς γίνεται αυτό. Το έχει συζητήσει το Συμβούλιο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος όσο γίνεται να περιορίζεται το κρατικό χρέος, το δημόσιο χρέος της χώρας. Για να ανακτήσουμε ή να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη των χρηματαγορών και να πέσουν τα επιτόκια. Για να μπορούν οι επιχειρηματίες των χωρών μας να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται. Όταν υπάρχει επιχειρηματικότητα, υπάρχουν και επενδύσεις και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Στη διαδικασία λοιπόν αυτή αμειώσουμε τα δημόσια χρέη, δεν έχουμε αυτόματα επενδύσεις. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση μόνο με οικονομίες και περίκοπες. Να πω και δύο λόγια για τη Λετωνία, τη χώρα μου. Τα τελευταία δύο χρόνια κατάφερε τα εξής. Ε, πρώτα έκανε πολύ σκληρή λιτότητα και εξοικονόμηση και φέτος το 1 τρίτο του προϋπολογισμού μας αφιερώθηκε σε δημόσιες επενδύσεις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα και λιτότητα και περικοπές αλλά και επενδύσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο κύριος Μαρινέσκου για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε ένα σημαντικό βήμα δημιουργώντας αυτόν τον μηχανισμό και ε, εγκρίνοντας τα μέσα ε, τα οποία θα επιτρέψουν αλλαγή των συνθήκων. Ε, με τον τρόπο αυτό θα δημιουργεί ένας συνεκτικός μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει σε περιόδους κρίσεως. Καλό βεβαίως είναι να έχουμε τέτοιους μηχανισμούς αλλά ακόμα καλύτερο να μην χρειάζεται να προστρέξουμε στον μηχανισμό αυτό η εφαρμογή ε, των αρχών της σωστής διακυβέρνησης μπορεί να αποτρέψει την ε, ε, χρήση του μηχανισμού αυτού. Συμφωνούμε με, το, με τη δημιουργία του Europlus και ελπίζουμε ότι ήταν και θεωρούμε ότι ήταν πολύ καλό και θετικό το ότι πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία συνέβαλε στην, στο, στο Europlus. Βεβαίως θα πρέπει να δημιουργήσουμε και νέες συνθήκες όσον αφορά ε, της, ε, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των, της εργατικής ε, δύναμης. Θεωρούμε ότι το μέλλον για να είναι λαμπρότερο θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστεί με την ενιαία αγορά, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να καλυφθούν οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούμε με την ε, ε, Κομισιόν όσον αφορά την πρόθεση της ε, πράξης για την ενιαία αγορά και οπωσδήποτε θα πρέπει να προωθηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να δοθεί λοιπόν όθηση στην ενιαία αγορά και φυσικά να υπάρχει πραγματικά ελεύθερη κυκλοφορία όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριος Μπουσουτήλ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αυτοί που προσπαθούν να φύγουν από τον πόλεμο της Λιβύης προσπαθούν αντίστοιχα να καταφύγουν ε, εις την Ευρώπη και επομένως εμείς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε ένα διτό φόβο. Ε, πρώτον δεν γνωρίζουμε για πόσους ανθρώπους μιλάμε, πόσοι είναι αυτοί που θα φτάσουν. Ο δεύτερος φόβος είναι ότι δεν ξέρουν και δεν ξέρουμε κατά πόσον η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει. Ε, είναι ένας φόβος τον οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί βεβαίως υπάρχει μηχανισμός αλληλεγγύης ο οποίος ε, υπάρχει ήδη στην Οδηγία 55 του 2001 πρέπει να χρησιμοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Μέχρι τώρα ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν το χρησιμοποιεί γιατί πρώτον δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Συμβούλιο ε, και θα ήθελα εδώ να κάνω έκκληση στον Επίτροπο Μπαρόζο ε, δηλαδή να μην υποβάλει αυτό το, αυτή την αιτιολογία δηλαδή από μόνη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ηγηθεί μιας προτάσεως έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Επίσης η Κομισιόν λέει ότι δεν έχουμε ε, ε, ε, τα, απαιτούμενα νούμερα. Ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως να διατυπώνουμε ένα τέτοιο, μια τέτοια άποψη γιατί τα νούμερα είναι εξαιρετικά μεγάλα για μια τόσο μικρή χώρα. Γι' αυτό λοιπόν καλώ τον πρόεδρο της Κομισιόν Μπαρόσο ε, να αρχίσει να εφαρμόζει τον, ε, κανονισμό, τον μηχανισμό αλληλεγγύης και ο, πρόεδρος, ο κ. επίσης να δείξει την απαραίτητη αλληλεγγύη. Για 1,5 λεπτό ο Πρόεδρε, νομίζω πως τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορεί πολιτικά και θεσμικά να κριθούν ικανοποιητικά. Το μήνυμα όμως της σημερινής συζήτησης, που είναι ότι η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί, είναι σημαντικό. Όπως είπε και ο πρόεδρος κ. Μπαρόσο, η οικονομική συγκυρία είναι αβέβαιη και δύσκολη. Ο συνάδελφος Φερχόσταφ μας επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βουλώσουμε κάποιες τρύπε, αλλά η κρίση ακόμα δεν έχει τελειώσει και ο πρόεδρος κύριος Βονρόμπα είπε πως κρεμούν προβλήματα. Έχουμε σφάλματα από το παρελθόν και έλλειψη των ενδεδειγμένων μέσων. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, να δούμε ποια είναι τα διδάγματα του παρελθόντος, να δούμε τι σημαίνει το υπερβολικό έλλειμμα και χρέος και πώς αυτά μας επιβαρύνουν. Γιατί είχα με πολιτικές των κρατών μελών και των θεσμών που είχαν αποτύχει και καλό θα ήταν να κάνουμε την ανάλυση αυτών και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και ελπίζω πως η νέα πράξη ενιαίας αγοράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι φιλόδοξη. Τουλάχιστον ε, το κεφάλαιο για το ψηφιακό τμήμα αυτής νομίζω ότι πλέον αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, αλλά όχι μικρή σημασία, είναι πως ε, σύντομα θα υπερψηφιστεί η νέα εστονική κυβέρνηση. Στις πρόφατες εκλογές οι ψηφοφόροι της ε, Εστονίας έδειξαν μία πολύ καλή ευρωπαϊκή συμπεριφορά γιατί υπερψήφισα μια κυβέρνηση που είχε κάνει σκληρές περικοπές και λιτότητα στη χώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία των αυθόρμητων τοποθετήσεων. Κάτσε Θέλω να σας ενημερώσω για την απόφαση που έλαβα για το τι μέλη γενέστε διαδικαστικά. Τουλάχιστον 20 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο βλέπετε ότι παρακάλεσα ήδη να αρχίσουν οι ψηφοφορίε στις 12 και 10 για να μπορέσουν να απαντήσουν οι κύριοι Μπαρόσο και Φαρόμπαϊ με τρόπο αξιοπρεπή χωρίς να τον ενοχλώνουν οι συνάδελφοι που θα εισέρχονται για να ψηφίσουν. Ταυτόχρονα σας προτείνω να ακούσουμε λίγο περισσότερους από τους μισούς, 12 με 13 συναδέλφους, 20 δεν προλαβαίνουμε σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θα δώσω πρώτα στο λόγο, το λόγο. Α, συγγνώμη. Να σας ενημερώσω για κάτι ακόμα, για να προσέχετε. Πάντα θα λέω ποιος έχει το λόγο και ποιος θα είναι ο επόμενος για να ετοιμάσετε, γιατί δεν έχετε κατάλογο μελητών. Τώρα, η κυρία Μαγκίνες πρώτη και στη συνέχεια ο κύριος Λάιχτφριτ. Ευχαριστώ πολύ Νομίζω ότι πολλά θετικά έχουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ατενίζοντας το μέλλον και νομίζω ότι σε σχέση με το παρελθόν και το ε, παρόν πήγαμε καλύτερα. Και βέβαια άκουσα τα όσα είπε η Κάθριν Ντέι στην Ιρλανδία την περασμένη εβδομάδα που μας είπε πως πια ε, δεν λάμπει το Ιρλανδικό θαύμα. Λοιπόν νομίζω ότι δεδομένων των τεστ αντοχής που έγιναν και της πολύ συνεκτικής και σφριγγυλής δράσης της νέας κυβέρνησης πιστεύω πως θα ξαναλάμψει το Ιρλανδικό θαύμα. Και αυτό το λέω για τον κόσμο που είναι σε κατάθλιψη, σε απογοήτευση και αισθάνονται ότι κουβαλάνε ένα πολύ βαρύ φορτίο που του έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για όσους αυτή τη στιγμή ε, καταλογίζουν κακή συμπεριφορά σε κράτη και σε λαούς θυμηθείτε πως πολλοί διασκέδασαν στο πάρτι που γινόταν και αναφέρομαι στις τράπεζες οι οποίες πέρασαν καλά πριν την κρίση. Εν πάση περιπτώσει έχουμε μια ηλιαχτίδα από το πρωί γιατί βλέπω πως ε, η, μετά τα τεστ αντοχής οι μεγάλοι παίκτες της παγκόσμιας οικονομίας στοιχηματίζουν υπέρ μας. Ελπίζω λοιπόν πως οι υπόλοιποι για τα επιτόκια θα μας κρίνουν με αλληλεγγύη. Αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε, ένα λεπτό έχετε στο ΚΑΤΣΔΙ. Αν θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα σε συναδέλφους σας να μιλήσουν, να τηρήσετε το χρόνο σας. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή, ακόμα αυστηρότερη. Ο κύριος Λάιφρυντ και μετά ο κύριος Οντζή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχω μερικές ερωτήσεις. Πρώτον, καλό είναι που επήλθε συμφωνία. Καλό είναι που η ευρωπαϊκή οικονομία και το ευρωπαϊκό νόμισμα τώρα προστατεύονται καλύτερα. Αλλά αρκεί και μόνη προστασία. Μήπως χρειάζεται να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, μήπως χρειάζεται να δώσουμε μια νέα ε, ορμή και όθηση ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία για να σώσουμε και αυτό που προστατεύουμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει ε, στην εξαγωγή ε, βοήου κρέατος και αγροτικών προϊόντων και όχι στη γνώση, στα πανεπιστήμια και αλλού. Όταν μας λέτε ότι το ταμείο είναι μείον, να κάνουμε μεταφορές πιστώσεων από εκεί που δίνουμε ε, χρήματα να τα μεταφέρουμε αλλού. Γιατί είναι πάντα οι ίδιοι αυτοί που επωφελούνται από αυτή την εκτρή κατάσταση. Γιατί κύριε Μπαρόσο εξακολουθείτε να αντιστέκεστε ε, και είστε κατά του φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Είστε με τις χρηματαγορές ή με τους πολίτες. Ο κύριος Σοντή και μετά ο κύριος Γκερέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προέδρους ε, των ομάδων που ακύρωσαν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις έτσι ώστε να συνεχίσει σύμφωνα με το άρθρο 15 η συζήτηση στην Ολομέλεια. Ο μηχανισμός σταθερότητας είναι κάτι καλό. Αλλά θα ήθελα να θέσω το ερώτημα του πολιτικού ελέγχου μετά και από αυτά που είπε και ο κύριος Λαμασούρ. Κυρίως δε το πρόβλημα της ρύθμισης αυτού του μηχανισμού. Να ξέρω, μάθω δηλαδή, ποιος θα δώσει την τελική ε, η απαλλαγή του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει ε, μια γενικότερη αναφορά ε, στο σύνολο των, ε, ροών, των οικονομικών ροών όσον αφορά τα ελλείμματα των κρατών. Επίσης, πιστεύω ότι η γενικότερη κατάσταση των δημοσίων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να την δούμε από κοντά γιατί λειτουργούν οι οίκοι αξιολόγησης με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ο κύριο Γκερέρο και μετά ο κύριο Βότσον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην αρχή τη παρέμβαση του ο κύριο Φαν Ρόμπαϊ μα είπε πω σε 49 μέρε είχαμε τρει συνόδου, τρία ευρωπαϊκά συμβούλια αποφασιστικά και μία σύνοδο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει κάτι το οποίο στο παρελθόν ήταν ένα γεγονός που γινόταν κάθε τρει μήνες. Έχει γίνει πια η σύνηθε τακτική για να κυβερνά κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανταποκρίνεται σε άμεσες προκλήσεις. Έχουμε λοιπόν και άλλες άμεσες προκλήσεις στον ορίζοντα, γιατί το μέλλον μας εξαρτάται από το πόσο ανταγωνιστική θα γίνουμε. Τι έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή για να δημιουργήσουμε γνώση. Λίγα από τα πανεπιστήμια μας είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Έχουμε ένα ποσοστό έρευνας και υπηρεσίας έρευνας που είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο των αναπτυγμένων χωρών και έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν ασχολούνται με τον κλάδο της έρευνας. Και για την ευρωπαϊκή διάσταση χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που θα συντονίζονται μεταξύ τους και προγράμματα τα οποία θα προκρίνουν την αριστεία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γότσον και στη συνέχεια ο κύριος Πάσκα. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι πρόεδροι της ε, ε, Κομισιόν και του Συμβουλίου μίλησαν για το Europlus και μετά για την ε, νέα αγορά. Θέλω να ρωτήσω τα εξής. Θα συμφωνήσετε με τον ε, πρόεδρο της ε, Κεντρικής Τράπεζας ε, ότι θα χρειαστεί ένας επιπλέον μηχανισμός και αν δεν συμφωνείτε αυτό συμβαίνει γιατί δύο αρμόδιοι δεν θέλουν να ομολογήσουν δημόσια αυτό που παραδέχονται ιδιωτικά. Δεύτερον, μια χώρα η οποία εφαρμόζει πραγματικά τους κανονισμούς 100% είναι η Νορβηγία και επομένως εδώ δεν μιλάμε απλώς για crash τεστ των ε, τραπεζών ή των εγκαταστάσεων, των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Μιλάμε για την ίδια την ελληνική τη Ευρώπης. Δεν πιστεύουν ε, οι αρμόδιοι πρόεδροι ότι δεν ήταν καλή η αλληλεγγύη που δείξαμε μέχρι τώρα. Ο κύριος Πάσκα και μετά ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Τα περισσότερα τα είπαν οι συνάδελφοι για το νέο μηχανισμό κρίσης της Ευρωζώνης. Μπορεί να βρήκαν λύση οι πρωθυπουργοί, αλλά θα πρέπει ακόμα να το συζητήσουν αυτό το θέμα με τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες στα κράτη-μέλη. Η κυρία Ραντίτσοβα ε, γύρισε από τις Βρυξέλλες και διαπίστωσε ότι στο κοινοβούλιο της χώρας δεν υπάρχει υποστήριξη θα πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός ελεγχόμενης χρεοκοπίας των αφαιρέγγιων κρατών. Και αυτό στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Ανταυτού χρησιμοποιείται το χρέος και αυξάνεται συνέχεια το χρέος. Αυτό δεν μπορεί κανένα υπεύθυνο κοινοβούλιο να το δεχτεί. Ακούστε και τους εμπειρογνώμονες της χώρας σας. Ο κύριος Μπρόνς και στη συνέχεια ο κύριος Κέλλη. 5 στο σημείο 5 της έκθεσης είπαμε πως θα έχουμε μέτρα πολιτικής για να ξεπεραστούν οι μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές στρεβλώσεις ή ε, επαναλαμβανόμενος και μιλάμε επίσης και για εμπορία με τρίτες χώρες. Νομίζω πως οι εισαγωγές από τις τρίτες χώρες και κυρίως από τις αναδυόμενες οικονομίες είναι ο βασικός λόγος που δημιουργεί ε, αυτή την ε, μη ανταγωνιστικότητα όπως επίσης και το, ε, την έλλειψη ισορροπίας στο εμπορικό ισοζύγιο. Λοιπόν, πώς θα του επιτρέψουν να κάνουν εξαγωγές χωρίς να κατεβάσουμε τους μισθούς στο επίπεδό τους. Όμως στη σελίδα 16 όταν μιλάμε για πρόσθεση ανταγωνιστικότητας υπονοείται κάτι τέτοιο που μιλάμε θα αξιολογηθεί η παραγωγικότητα, η εξέλιξη των μισθών και θα προσαρμοστούν οι ανταγωνιστικές μας ανάγκες. Τι σημαίνει αυτό. Ένα και μόνο. Μείωση, εξίσωση προς τα κάτω των μισθών έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας με αυτά των αναδειωμένων αγορών όπου το ελεύθερο εμπόριο βέβαια αποτελεί μια ιερή αγελάδα, αλλά εκεί θα πρέπει να τοποθετήσουμε και τους μισθούς του Ευρωπαίου εργαζομένου. Ο κύριος Κέλλη και μετά ο κύριος Ταραμπέλα. Δεν θέλω να ε, ε, ε, υποχρεώνω κάποιον να κάνει κάτι και το ίδιο δεν θέλουν και οι Ιρλανδοί. Οι Ιρλανδοί προσπάθησαν πάρα πολύ έτσι ώστε να αποφύγουν την χρεοκοπία. Αλλά βεβαίως οι υπεύθυνοι σαφώς δεν είναι οι πολίτες της Ιρλανδίας. Είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα των τραπεζών και των κυβερνήσεων. Ζητούμε λοιπόν μείωση των επιτοκίων πρώτα απ' όλα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, την Επιτροπή και τον Πρόεδρο Μπαρόζο προς, κατά αυτή την έννοια. Δεύτερον, πιστεύουμε όντως ότι θα πρέπει να πληρωθεί κάποιο τίμημα ε, και θα πρέπει να... Ε, αλλά το τίμημα αυτό αν, ε, θα πρέπει να μειωθεί, να υπάρχει ένα κούρεμα ή εν πάση περιπτώσει ένα σημάζεμα αυτού του χρέους. Εάν αυτά τα δύο πράγματα συμβούν τότε πραγματικά δεν θα χρεοκοπήσουμε, θα ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Ο κύριος Ταραμπέλα και με τον κύριο Σταμπάιντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. μας ε, ε, νομίζουμε ότι με το Europlus ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας της Ευρώπης ε, όπου θα δημιουργηθούν μια σειρά προβλημάτων κατέβασμα των μισθών, μείωση της αγοραστικής αξίας, μεγαλύτερη ηλικία συνταξιοδότησης κλπ. κλπ. Φοβούμε ότι το Συμβούλιο δεν έμαθε τα μαθήματα της κρίσης βεβαίως θέλουμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική δημοσιονομικής αυστηρότητας και πειθαρχίας, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να στηγυρίσουμε την πλάτη μας στους πολίτες που είναι η μόνη μας ελπίδα διαφυγής από την κρίση αυτή. Ε, ξεχνάτε ότι ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει και αυτός να φέρει ένα μερίδιο της ευθύνης, συγγνώμη, θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει μια και φέρει ένα μεγάλο ε, τμήμα ε, της ευθύνης. Το Συμβούλιο τελικά το μόνο που αποφασίζει κερδίζει είναι ε, να πληρώνει όχι το κεφάλαιο αλλά μονάχα οι πολίτες και αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταμπάιτη. Και μετά ο κύριος Όμπαμαϊ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος, ο πρόεδρος Βαν Ρόμπεϊ αναφέρθηκε στη συμφωνία Europlus και θεώρησε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια νέα φάση συντονισμού των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, ο οποίος είναι και προεδρεύον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως, αναφέρθηκε σε ένα νέο πυλώνα του Ευρωπαϊκού Συστήματος. Δυστυχώς το όνομα της Ουγγαρίας όμως δεν αναφέρεται στον κατάλληλο διάλογο που ανέφερε ο Πρόεδρος Βον Ρόμποϊ, διότι δυστυχώς δεν, δεν ε, συμμετέχει η Ουγγαρία ε, στη Συμφωνία Europlus. Πολλοί ε, εμπειρογνώμονες, οικονομολόγοι Ούγγροι και οι πολίτες της Ουγγαρίας δεν κατανοούν αυτήν την συμπεριφορά. Η Ουγγαρία όμως είναι μια μικρή ανοιχτή οικονομία και ε, επίσης με την εναρμόνιση ε, της φορολογητέας βάσης ε, θα είναι μεγαλύτερος και ο φορολογικός ανταγωνισμός. Είναι κρίμα πάντως. και μετά η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταθλήτρια τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, φίλοι του Καντάφη, φίλοι της πυρηνικής ενέργειας. Όλα αυτά έχουν καταρρεύσει. Μετά την Ελλάδα τώρα και η Πορτογαλία ε, ε, υποβαθμίζεται από τους οίκους αξιολόγησης και οι τράπεζες και οι διάφοροι κερδοσκόποι τώρα ποντάρουν στη χρεοκοπία κρατών. Πού είναι τα ευρωομόλογα. αν θα παραμείνουν οι ε, υποχρεοκοπία χώρες στην Ευρωζώνη είναι αρχή και το τέλος του ευρώ. Έχουμε τώρα ε, ρεύματα προσφύγων από την ε, Αφρική. Δεν θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ορθοποδήσουν στις χώρες τους. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την πυρηνική ενέργεια και να χρησιμοποιούμε καλύτερα τους οικονομικούς μας πόρους παρά σε αυτό το καζίνο το διεθνώς των οίκων αξιολόγησης. Ευχαριστώ η κυρία Γκόμες και μετά η κυρία Μπένοβα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή πιέζεται η Πορτογαλία να δεχτεί βοήθεια. Εμεί δεν θέλουμε βοήθεια, γιατί αυτό προσπαθούν να κάνουν είναι να μα βυθίσουν και να βυθίσουν το ευρώ. Στην Ευρώπη λοιπόν τη αλληλεγγύη, τη κοινωνική διαχείριση, όλα αυτά έχουν γίνει μάταια και άδεια λόγια οι τράπεζες προσπαθούν να μας πιέσουν μέσα σε μια δίνη χρέους στην οποία προσπαθούν να μας βυθίσουν. Τώρα για το Europlus που υποτίθεται θα μας βοηθήσει στο να ανακάμψει η οικονομία μας και να αναπτυχθεί ε, η χώρα και να έχουμε περισσότερη απασχόληση, να σας πω πως όλα αυτά δεν θα μας βοηθήσουν. Έχουμε πολύ μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη, οι οποίες δεν καταραίουν και αντί να καταρρεύσουν οι τράπεζες, καταραίουν τα κράτη-μέλη. Μόνο η ύπαρξη συμφερόντων μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο εξακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο να στηρίζουν τους φορολογικούς παραδείσους Λοιπόν, θα πρέπει αυτές τις μαύρες τρύπες ε, που δεν τολμά να θίξει κανείς, εμείς να τις φωτίσουμε. Η κυρία Μπένοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι, καταρχάς θα ήθελα να ε, σας επιστήσω την προσοχή ε, στη λάθος εστίαση της απόφασης από τη μια ανάπτυξη, από την άλλη περικοπές. Πώς θα γίνει αυτό. Εμείς θα πρέπει να ενισχύσουμε την απασχόληση και τη μεγέθυνση της οικονομίας. Ε, αλλιώς θα πληρώσουν την κρίση οι πολίτες. Χάνουν έτσι κι αλλιώς τις θέσεις τους και μετά υφίστανται και τις περικοπές ε, των κυβερνήσεων. Σε τελική ανάλυση τα πληρώνουν όλα οι φορολογούμενοι πολίτες. και δεν συμμετέχουν εκείνοι που κερδοσκοπούν εις βάρος ε, του ευρώ. Αυτό που χρειάζεται είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, η διάσωση του ευρώ και να συμμετέχει παρακαλώ και η ιδιωτική οικονομία. Η κυρία Βέρτμαν και τελευταίο στη συζήτηση ο κύριος Μπαλτσίτης. Η κυρία Βέρτμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με την αλλαγή της συνθήκης, ο μόνιμος ε, μηχανισμός ε, έχει δρομολογηθεί. Παρακαλώ όλους να τηρήσουν τα κριτήρια. Γιατί αν έρθει και άλλη χώρα σε αυτή την κατάσταση, η κρίση διαρθρωτική ε, γίνεται πλέον ανεύθυνη θα πρέπει όλες οι χώρες να τηρούν τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις και να υποχρεώνονται να κάνουν οικονομίες. Μόνο έτσι θα λειτουργήσει το σύστημα. Μας έδειξε η κρίση στην οικονομία πόσο ασφαλής μπορεί να είναι η πυρηνική ενέργεια. Η φύση είναι πιο ισχυρή από τον άνθρωπο. Τεστ αντοχής θα πρέπει ε, να γίνουν με μεγαλύτερη ε, προσοχή ε, και να σταματήσουν τα πυρηνικά εργοστάσια. Το είδαμε και στο Τσέρνομπιλ. Επιτέλους να επικεντρωθούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ. Τελευταίο στη συζήτηση αυτή ο κύριος Μπαλτσίτης, ε, λεπτό, μια στιγμή, και μετά θα έχουμε δώσει το λόγο σε 15 συναδέλφους, αντί σε 5, όπως προβλέπετε. Δυστυχώς παραπάνω δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ο κύριος Μπαλτσίτης τελευταίος στο ΚΑΤΣΙΑΙ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Είναι καλό που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τελικά κατάφερε να συμφωνήσει πάνω σε πολύ σημαντικά θέματα ε, και ε, η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει βεβαίως ε, να ε, ε, δοθεί βάση στην δημοσιονομική πειθαρχία των χωρών, καθώς επίσης και στην πρόθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί σημασία στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής 2020 και βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη εποπτεία των δράσεων των κρατών ε, μελών και τα προγράμματα ε, υλοποίησης, σύγκλησης και σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε από κοντά να κοιτάξουν την κατάσταση των οίκων αξιολόγησης. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν η διαδικασία αυτή και η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπαρόσο, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Όσον αφορά την αξιολόγηση του τελευταίου Συμβουλίου, νομίζω ότι η ανάλυση την οποία σας υπέβαλε ήταν μάλλον ισορροπημένη ε, και μάλλον λογική. Πιστεύω ότι είναι ορθό να αναγνωρίσουμε ότι έγιναν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την ίδια τη δομή. Τώρα, εάν συγκρίνουμε με αυτά που δεν είχαμε στο παρελθόν, οπωσδήποτε η πρόοδος είναι σημαντική. Ας πούμε, η δημιουργία ενός ε, μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας που δεν προεβλέπεται από την συνθήκη και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε στην δημιουργία ενός εργαλείου που δεν υπήρχε πριν. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινεί στην αξιολόγησή μας και να διαπιστώσουμε ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος ε, όσον αφορά την ανταπόκριση στην κρίση και όσον αφορά την δυνατότητα αντιμετώπισης των ανεπαρκειών του παρελθόντος ε, όσον αφορά και τους μηχανισμούς αλλά και τις πολιτικές. Ταυτοχρόνως όμως το λέω και το λέω σαφώς ότι ενδεχομένω αυτές οι κινήσεις δεν είναι αρκετές. Ε, ένα πράγμα είναι να έχει κανείς μία δομή και ένα πλαίσιο, ένα περίβλημα και ένα άλλο είναι να το γεμίσει με συγκεκριμένες στρατηγικές. Θα δούμε λοιπόν, δημιουργούμε ένα μηχανισμό και θα δούμε τι μπορούν να κάνουν τα θεσμικά όργανα και οι κυβερνήσει όσον αφορά την ουσία την οποία θα δώσουν σε αυτά τα εργαλεία, γιατί η ουσία υπερέχει των μηχανισμών και των εργαλείων. Πιστεύω ότι όσον αφορά τη διαφάνεια ήμουν αρκετά ε, ε σαφή. Η Κομισιόν βεβαίω θα είχε προτιμήσει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Υπογραμμίσαμε, α πούμε, ότι όσον αφορά τον μόνιμο μηχανισμό σταθερότητα, ε, εμείς θέλαμε περισσότερη ευελιξία όμως δεν κατέστη δυνατή συνένεση σε αυτήν την μεγαλύτερη φιλοδοξία. Απ' την άλλη πλευρά θεωρώ ότι δεν είναι ορθό να απορρίψουμε όλα αυτά τα οποία επιτύχαμε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι σημαντικό γιατί μερικοί υπονόησαν ότι η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει και άλλες προτάσεις. Κοιτάξτε, όλες αυτές τις προτάσεις που εσείς αναφέρατε τις έχει ήδη κάνει η Κομισιόν. Την 9η ε, Μαΐου του 2010 και εγώ ίδιος ε, και ο Επίτροπος Ρένα υποβάλαμε νομοθετικού περιεχομένου πρόταση όσον αφορά την κοινωτική προσέγγιση του μηχανισμού σταθερότητας. Προτείναμε την αμοιβαιότητα όσον αφορά την διαχείριση του κινδύνου, joint and several guarantees. Όμως απερίφθη αυτό από τα κράτη-μέλη απερίφθη. Όχι από εσά. Ναι, εντάξει, το δικό σα όχι. Μα κύριε Φερχόφστατ, τι να σα πω. Παρατηρήσει εκτό μικροφώνου του κύριου Φερχόφστατ. Μπορώ να σας πω ότι εμείς υποβάλαμε το κείμενο στην ε, διάσκεψη ορυφής της Ευρωζώνης και απερίφθη από μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά ε, το συγκεκριμένο θέμα ε, της ομοφωνίας και της ε, ε, ψήφου κατά πλειοψηφίας. Εγώ το πρότεινα. Το πρότεινα την παρουσία του ε, Προέδρου Φαν Ρόμπεϊ ε, ε, έτσι ώστε να δεχτούν την ενισχυμένη πλειοψηφία τα κρατημέλη αλλά απερίφθη η πρόταση μπορούμε να το υποβάλουμε, να ξαναπροτείνουμε και να επιμείνουμε αλλά κοιτάξτε τουλάχιστον να μην κάνετε λάθος παραλήπτη των ετοιμάτων σας να στρέφεστε προς αυτόν που πρέπει να στραφείτε για να ρωτήσετε τα, ε, ζητήματα αυτά και βεβαίω συμφωνώ ότι θα πρέπει ε, όσον αφορά τα ευρωομόλογα να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Εδώ και 30 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για ευρωομόλογα αλλά κανείς, ε, μάλλον όχι κανείς, αλλά πολλές χώρες δεν τα δέχτηκαν. Ενδεχομένως τώρα λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε project bonds για συγκεκριμένη χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Θα δούμε, θα δούμε όταν θα κάνουμε την πρόταση, θα δούμε ποιο θα συμφωνήσει με αυτήν την προσέγγιση ε, των ευρωπαϊκών επενδύσεων και ενδεχομένω, εσείς μπορείτε μέσω πιέσεως των δικών σα κομμάτων ε, να ε, διασφαλίσετε στήριξη αυτών των δημοσιονομικών προοπτικών και εκεί ίσως θα μπορέσουμε να δουλεύουμε δουλέψουμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτές είναι, ε, οι, φιλοδοξίε Αυτές είναι οι φιλοδοξίες μας όσον αφορά το ζήτημα. Τώρα, τα κοινωνικά ζητήματα. Πρέπει να σας πω ότι αγωνίστηκε πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε στη στρατηγική 2020 να υπάρχει μεγαλύτερη υπογράμμιση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων. Δεν ήταν πολύ εύκολο γιατί πολλοί ηγέτες έλεγαν ότι βάσει της αρχής επικουρικότητας δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει άμεση δράση όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα και όσον αφορά την εκπαίδευση. Ας προσπαθήσουμε τώρα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 όπου υπήρχε η δυνατότητα ε, να υπάρξει κάποια συνένεση έτσι ώστε ε, να ε, ε, βάλουμε στη στρατηγική αυτή την καταπολέμηση της ένδυας ας πούμε ε, να, να, να βάλουμε και κάποια στοιχεία επίσης για επενδύσεις στην γενοτομία και στην εκπαίδευση πρέπει να σας πω όμως επιτρέψτε μου δηλαδή να σας πω το εξής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πριν από λίγο καιρό, νομίζω πριν από δύο χρόνια αν δεν κάνω λάθος, υπέβαλε λοιπόν κάποιες προτάσεις να υπάρξει επίγουσα διατροφική βοήθεια σε κάποιες χώρες γιατί και στην Ευρώπη είναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, δεν, ε, ε, δεν καλύπτουν την πείνα τους. Ε, υπάρχουν προβλήματα όχι μονάχα σε αναπτυσσόμενες χώρες ε, αλλά ε, και στην Ευρώπη και φτάσαμε τελικά να μας σύρουν στην, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί ζητούσαμε ένα μηχανισμό στήριξης των φτωχών ανθρώπων που δεν καταφέρνουν να τραφούν όσο πρέπει. Αυτή είναι η κατάσταση. Βεβαίως εμείς θέλουμε πιο ισόρροπη ανάπτυξη, πιο δίκαιη η ανάπτυξη. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μας στηρίξει και το Κοινοβούλιο και τα, να μας στηρίξουν και τα κράτη-μέλη στις προτάσεις μας αυτές. Και επομένως νομίζω ότι ε, λανθάνουμε στόχο όταν στρεφόμαστε μονάχα ε, εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή η οποία έκανε ε, πρώτη τις πιο κοινωνικές, τις πιο δίκαιες προτάσεις και ήταν πάντα και από την αρχή υπέρ της ορθότερης οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι, ε, λέμε, πρόβλημα της Ευρώπης. Λες και καμία κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη γιατί άφησε το χρέος της να φτάσει σε τέτοια επίπεδα ή ε, γιατί οι τράπεζες είχαν ανάπτυξη πολλές φορές πάνω από το ε, ΑΕΠ. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ελληνικής, αλλά ε, βεβαίως ε, και απαντήσεις όσον αφορά τις ευθύνες που έχει ο καθένας. Εγώ είμαι, υπε, ε, ε, υπερήφανος σαν πρόεδρος της Επιτροπής, ε, γιατί εμείς προσπαθήσαμε πολύ έτσι ώστε να μειωθεί το επιτόκιο χρέος που πληρώνει η Ελλάδα, δανεισμού που πληρώνει η Ελλάδα και προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο και για την Ιρλανδία και ε, ξέρουμε ότι και οι Έλληνες ε, πολίτες και οι Ιρλανδοί περνάνε πάρα πολύ δύσκολες ώρες ε, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει και θα πρέπει να, ενεργήσουμε με τρόπο ώστε το χρέος να είναι βιώσιμο. Μαζί πρέπει να βρούμε κοινέ λύσεις έτσι ώστε να αποφύγουμε κάτι που ανέφεραν πολύ μεταξύ ημών, το πρόβλημα κάποιου ε, μοιράσματο της Ευρώπης, κυρίως ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο, το κέντρο και την περιφέρεια και μένα με φοβίζει αυτό. Θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν έχουμε Ευρώπη πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, έχουμε μία και μοναδική Ευρώπη, μία Ευρώπη στην οποία μπορούν να βλέπουν τον εαυτό τους όλοι οι πολίτες. Τώρα για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πρέπει να σου το πω πως εγώ το κείμενο αυτό και στην ομάδα των 20 στην G20 το υπερασπίστηκα ε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το απέρριψε ένα τεράστιο κομμάτι των εταίρων μας στην ομάδα των 20. Το θέμα είναι κατά πόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμεί μπορούμε ή όχι, θα έπρεπε ή όχι να έχουμε τέτοιο είδος φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ας είμαστε ειλικρινείς. Είναι αρκετά τα κράτη-μέλη τα οποία είναι κάθετα αντίθετα με την εισαγωγή του φόρου αυτού και δεν πρόκειται να συμφωνήσουν. Στην τελευταία σύνοδο το είπα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτή τη στιγμή μια μελέτη αντικτύπου σε όλον το χρηματοπιστωτικό κλάδο και θα κατεβάσουμε προτάσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι ανακοίνωσε στο Συμβούλιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί τουλάχιστον στα συμπεράσματα του Συμβουλίου έχουμε αναλάβει έχουμε βρει τη δέσμευση να εξεταστούν οι προτάσεις τις οποίες θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το φόρο αυτό γιατί πιστεύω πως είναι θέμα δικαιοσύνης είναι να πούμε στο χρηματοπιστωτικό κλάδο ο οποίος σε κάποιο βαθμό είναι υπεύθυνο για την κρίση αυτή να ζητήσουμε να ζητήσουμε για να είμαστε δίκαιοι κάποια βοήθεια για να ξεπεράσουμε την κρίση. Και οι προτάσεις αυτές θα κατατεθούν, επαναλαμβάνω, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το CCTV επίσης έχουμε αντίθεση από κάποιους στο Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως έχει καταθέσει και εκεί προτάσεις και θα τις υπερασπιστούμε γιατί θεωρούμε πως είναι σημαντικό κάτι τέτοιο για να ε, ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά, η ενιαία αγορά. Άρα λοιπόν αυτή είναι η θέση μας. Άρα λοιπόν αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου έχουμε συζητήσει διαδικασίες και μέσα και το κάνουμε για πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούν τα μέσα αυτά και οι διαδικασίες αυτές να μας εξυπηρετήσουν επί της ουσίας. Γιατί είναι η ουσία το βασικό. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το τάδε μέσος υποκατάστατο της ουσιαστικής πρόοδο που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνη για να θέλει κανεί να επενδύσει στις χώρε μα. Και πώ θα το αποκτήσουμε. Θα πρέπει να είμαστε πιο βιώσιμοι, πιο ανταγωνιστικοί, ε, πιο καινοτόμοι. Οι επενδύσεις θα προσελκυθούν εάν εφαρμόσουμε την Ευρώπη του 2020 γρήγορα και με επιτυχία. Εάν επιδιώξουμε τους στόχους μας. Εάν αποκτήσουμε μια Ευρώπη η οποία είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη. Μέσα στο πνεύμα τη Αλληλεγγύη, γιατί και στην αλληλεγγύη θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα κράτη-μέλη. Και εκεί συμπεριλαμβάνω και την Πορτογαλία. Και επειδή ακούστηκε μια ερώτηση για την Πορτογαλία, ο φίλο μου Μάρτιν Σούλτ πρέπει να σου πω φίλε Μάρτιν πω εγώ ω πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν πρόκειται να παρέμβω στην εσωτερική πολιτική τη Πορτογαλία. Εάν κάποια μέρα εσείς πλέον δεν είστε πρόεδρος σοσιαλιστικής ομάδας και έχετε κάποια άλλη θύση, νομίζω πως στη νέα αυτή θέση που θα έχετε ε, θα ε, κάνετε τη δουλειά σας χωρίς να παρεμβαίνετε με τα όσα συμβαίνουν στη σοσιαλιστική ομάδα αφού δεν θα είστε πια εκεί. Λοιπόν, η πολιτική κρίση στην Πορτογαλία δεν διευκόλυνε την κατάσταση. Η Πορτογαλία ήδη ήταν σε αρκετά δύσκολη θέση. Όμως εμείς, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, θα πρέπει να σεβαστούμε την εθνική δημοκρατία, τις αποφάσεις του Εθνικού Κοινοβουλίου και να, να περιμένουμε τώρα το τι θα γίνει γιατί οι Πορτογάλοι θα δώσουν την απάντηση. Λοιπόν, εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξουμε τους Πορτογάλους να βρουν την βέλτιστη λύση στα πλαίσια βέβαια του σεβασμού των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Πορτογαλία. ενώπιον των Ευρωπαίων εταίρων της. Μέσα στο πνεύμα αυτό η δραστήρια και ενεργή αλληλεγγύη που θα δείξουμε θα μας βοηθήσουν να δώσουμε μια απόκριση στην κρίση. Σήμερα η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε είναι πως είστε μάλλον απεσιόδοξοι εδώ. Βέβαια, εσείς εκπροσωπείτε, στη αιρετή εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Και όντω αυτή τη στιγμή αυτό που μα μεταφέρετε είναι αυτή την απεσιοδοξία που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Είμαστε ανήσυχοι, αλλά θα πρέπει να σταθούμε, να βρούμε την τόλμη, την πολιτική τόλμη και το καθαρό μυαλό που θα μας επιτρέψουν να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Δεν θα πρέπει να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη με ενθουσιασμό δίπλα σας, δίπλα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δίπλα σε όλους τους θεσμούς να δώσει τη μάχη για μια πιο βιώσιμη, πιο δίκαιη, πιο ίση και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Thank you. Thank you much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν δεχόμαστε γαλάζιες κάρτες. Τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Λοιπόν, μιλώ αγγλικά, δεν έχετε ακουστικά, όλοι καταλαβαίνετε αγγλικά. Βλέπετε ότι η ψηφοφορία θα αρχίσει μόλις στις 12 και 10. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε ησυχία γιατί θέλουμε να ακούσουμε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Και να έχει την προσοχή σας. Ίσως να μην με τόσο κύριε Φαν Ρομπέ όπως ο κύριος Μπαρόσο, πάντως έχετε το λόγο. Μια στιγμή παρακαλώ. E? Καθίστε. Καθίστε παρακαλώ και εσείς στο ΕΛΚ. Καθίστε. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ καθίστε. Δεν θέλω να μιλάτε μεταξύ σας, μόνο εκτός εθούσης. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να λάβει το λόγο τώρα είναι ο κύριος Φαν Ρομπέι. Κύρια Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που μπορώ να απευθυνθώ σε ένα τόσο τεράστιο ακροατήριο. Είναι ίσω οι περισσότεροι ευρωβουλευτέ που με ακούν από τότε που έγινα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νομίζω πως μάλλον δεν ήρθατε μόνο για μένα, δεν ήρθατε μόνο για να με ακούσατε στην αίθουσα. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για όλες τις παρατηρήσεις που κάνατε και για αυτά τα σχόλια τα οποία ήταν θετικά και για αυτά τα οποία ήταν αρνητικά, για όλα όσα μας είπατε. Και πρέπει να σας πω πως αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι πως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ομοφωνία. Και αυτή η ομοφωνία μας οδηγεί στο να συμφωνήσουμε με όλους τους ε, συναδέλφους σας από οποιοδήποτε κόμμα και να προέρχονται, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Έχουμε συντηρητικούς, ε, ε, φιλελεύθερους, σοσιαλιστές, όλοι οι οποίοι ανήκουν στις δικές σας πολιτικές οικογένειες και κάθε φορά το προσπαθούμε και νομίζω τα καταφέρνουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Μας είπατε προηγουμένως πως θα πρέπει να είμαι ο ιδεαλιστής ε, που εξυπηρετεί τις ανάγκες μας ο δημιουργός ονείρων. Όχι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Και τι κάνω. Στο μέτρο του δυνατού βέβαια και νομίζω πως εδώ έχω και μάρτυρο να με στηρίξει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι να ενεργώ έτσι ώστε στις περισσότερες περιπτώσεις να έχουμε μία σύγκληση μεταξύ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και θα σας δώσω το παράδειγμα. Έχουμε μία task force. Ήμασταν πολύ κοντά, ήμασταν πολύ κοντά για την οικονομική διακυβέρνηση και για την σχετική task force να βασιστούμε στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συμφωνήσουμε και θα το δοκιμάσουμε, θα το προσπαθήσουμε μαζί με εσά, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις προτάσεις. Ο ρόλος, μας, ο ρόλος μου είναι λοιπόν του αναζητητή της συνένεσης η οποία θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοινοτική στη φύση της και ελπίζω να κρίνετε κι εσείς θετικά στις προσπάθειες που έχω να κάνω για το σύμφωνο Europe Plus. Ξέρετε, πως είχαμε ένα μικρό έγγραφο το οποίο ήταν η αρχή της συζήτησης και είναι το έγγραφο από το οποίο προέκυψε αυτό το σύμφωνο. Οι περισσότεροι εσείς μας είπατε πως θέλετε η χώρα σας να υπογράψει το σύμφωνο αυτό και να συμμετάχει σε αυτό. Άρα λοιπόν είναι ένα κείμενο το οποίο δεν είναι και τόσο άσχημα αν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή. Καταφέραμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι αρκετά φιλόδοξο έτσι ώστε οι οικονομίες μας να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να είναι βιώσιμες οι δημόσιες δαπάνες και η εκτέλεση σε εθνικό επίπεδο, γιατί μιλάμε τώρα για εθνικές αποφάσεις, να γίνεται με έναν σχετικά κοινό τρόπο. Ε, κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, ζητώ από την αίθουσα περισσότερο ησυχία. Σας παρακαλώ πολύ στα αριστερά της αίθουσας, καθίστε. Και σας παρακαλώ πολύ μη μιλάτε μεταξύ σας. Κύριε Σρέντερ, παρακαλώ καθίστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να συνεχίσετε κύριε Φαν Ρόμπαϊ. Λοιπόν, μην νομίζετε, μην νομίζετε πως θεωρώ πως είναι όλοι εδώ για μένα, κυρία Πρόεδρε. Προσπαθώ να σας διευκολύνω τη ζωή. Αν δεν το επιθυμείτε, στο μέλλον δεν θα το ξανακάνω, κύριε Πρόεδρε. Η δεύτερη μου παρατήρηση σχετίζεται με τη μεθοδολογία, κατά κάποιο τρόπο. Ακούστηκαν πάρα πολλά επικριτικά σχόλια προς την Ευρώπη και πολλές φορές δικαιολογούνται επί της ουσίας, αλλά δυστυχώς δεν συμφωνούν με τα όσα έχουμε στις συνθήκες. Για παράδειγμα, πυρηνική πολιτική, το ενεργειακό μείγμα, εθνική αρμοδιότητα. Ναι, είναι εθνική αρμοδιότητα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εκεί. Όμως για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών Πρέπει να σας πω πως σε μεγάλο βαθμό και αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Υπάρχουν όμως κοινοτικέ αρμοδιότητες, ευρωπαϊκές αρμοδιότητες και εκεί. Προσπαθήσαμε λοιπόν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να τις προκρίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιο ρόλο να παίξει εδώ μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τόσο αποφασίστηκαν πριν από ορισμένε μέρε. Θα πρέπει όμω εμεί να λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο των συνθήκων. Μιλήσαμε για του ελάχιστου μισθούς. Μιλήσαμε για αβεβαιότητα, για κοινωνική αδικία. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις όλα αυτά έχουν να κάνουν με εθνικά μέτρα. Πρέπει να προσθέσω εδώ πως αρκετά από τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν στο μέλλον για τα δημόσια, τις δημόσιες δαπάνες είναι μέτρα όπου οι εθνικές αρχές θα πάρουν ακόμα και χωρίς να τις πιέσει η Ευρώπη. Εμείς τι κάνουμε. Πιέζουμε επιπλέον. Γιατί έχουμε ένα ευρωπαϊκό νόμισμα το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Τα μέτρα λοιπόν τα οποία πρέπει να πάρετε στις χώρες σας είναι μέτρα τα οποία είναι για το δικό σας συμφέρον, σε εθνικό επίπεδο, για να εξασφαλίσετε το μέλλον της δικής σας χώρας. Αυτό που κάνει η Ευρώπη είναι να προσθέτει μία επιπλέον πίεση προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Μην καταδικάζετε και κατηγορείτε άδικα την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά τα μέτρα. Τώρα για τη διακυβέρνηση, την οικονομική διακυβέρνηση θα εργαστούμε ακόμα περισσότερα. Εμείς θα συνεργαστούμε ως Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιώσουμε το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης και όπως και σε άλλες περιπτώσεις είμαι πεπισμένος πως θα βρούμε μία συμβιβαστική λύση. Ίσως να έχουμε τον διοικητή μιας ε, κεντρικής τράπεζας 17 ε, κρατών ε, μελών ο οποίος θα μπορεί να ε, με συγχωρείτε, ίσως έχουμε έναν από τους 17 διοικητέ κεντρικών τραπεζών που πέραψαν το σύμφωνο που στάθηκε πάρα πολύ επικριτικά στο σημείο αυτό. Οι υπόλοιποι όμως πρέπει να σας πω πως ήταν μάλλον θετικοί και αν σας ενδιαφέρει μπορώ να σας δώσω και το όνομα και να σας πω ακριβώς τι υπόθηκε αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο για την τρέχουσα κρίση. Ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον, ξέρουμε ποια είναι τα μέσα τα οποία εγκρίναμε, σημαντικές αποφάσεις, αλλά έχουμε και το παρελθόν. Και πρέπει να σας πω πως πρέπει να διαχειριστούμε τα όσα έγιναν στο παρελθόν. Γιατί Ακόμα και με τους μηχανισμούς διευκόλυνσης, σταθερότητας, με την οικονομική διακυβέρνηση, με το σύμφωνο, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των τραπεζών που πιέζονται από τις αγορές. Άρα λοιπόν έχουμε αφενός το μέλλον για το οποίο κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά και το παρελθόν, όπου είχαμε μια έλλειψη πολιτικών σε κάποια κράτη-μέλη και έχουμε και μία έλλειψη πολιτικών στο παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας το πούμε ανοιχτά, ας δούμε και τις δικές μας ευθύνες. Θα το κάνουμε. Λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα και με τον τρόπο αυτό η κρίση δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Αλλά θα πρέπει να διαχειριστούμε εντωμεταξύ όπως σας είπα και τα διδάγματα και τα ίχνη που άφησε επάνω μας το παρελθόν. Για κάποιες χώρες τις οποίες γνωρίζετε και οι οποίες είναι στα πλαίσια κάποιου προγράμματος όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα και κάποια άλλα κράτη για τα οποία θα λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να μην ενταχθούν ενδεχομένω αυτά τα προγράμματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τα μέτρα αυτά πριν από ένα χρόνο. Όχι. Υπήρξαν σημαντικά λάθη στο παρελθόν. Δυναμητίστηκε πριν από 7-8 χρόνια το σύστημα ε, σταθερότητας γιατί διαφορετικά και αν δεν το είχαμε κάνει αυτό θα είχαμε πολύ πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να αποφύγουμε τις κρίσεις. Η οικονομική ανάπτυξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, από το 2010 έχουμε ένα μέσο όρο ανάπτυξης 2%. Είναι ο μέσος όρος της δεκαετίας 1999-2008. Ε, από το 2010 λοιπόν και στο 2011 έχουμε μέσο όρο ανάπτυξης 2%. Πρέπει να ε, ε, πάμε καλύτερα, μα βεβαίως πρέπει να πάμε. Τα δημόσια εργαλεία είναι τα μόνα, οι μόνες δυνατότητες. Μα βεβαίως και όχι. Η ενιαία εσωτερική αγορά είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, θα πρέπει να την εμβαθύνουμε. Υπάρχουν επ' αυτού προτάσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα τι ξανασυζητήσουμε μετά από μερικέ εβδομάδες στο Συμβούλιο του Ιουνίου και βεβαίω και το φθινόπωρο θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Τέλος, για την Λιβύη μπορεί κανείς να είναι πολύ επικριτικός. Όμως, χωρίς την Ευρώπη θα είχαμε ε, δει σφαγές και λουτρό αίματος σε την ε, Λιβύη. Χωρίς την ευρωπαϊκή ηγεσία θα είχαμε σφαγές. Είναι γεγονός ότι πολλοί μεταξύ ημών είσαστε πολύ επικριτικοί απέναντι στην Ευρώπη, όμως έγκαιρα ε, δράσαμε και χωρίς την Ευρώπη τίποτα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει σε επίπεδο διεθνές αλλά και Ηνωμένων Εθνών και ό,τι κι αν πει κανεί, νομίζω ότι θα πρέπει να, να παραδεχτεί τελικά την αλήθεια. Αμαρτήσαμε κατά το παρελθόν. Ναι, είχαμε σωστές πολιτικές. Όχι. Διορθωθήκαμε. Ναι. Ε, και ε, ε, νομίζω ότι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει τα εύσημα της διόρθωσης. Και να τελειώσω με κάποια λόγια στη γλώσσα μου. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Έπινγκ που ήταν απογοητευμένος. Εγώ να δείτε πόσο είμαι απογοητευμένος από την έλλειψη πνευματικής ειλικρίνειας. Από την ειλικρίνειά σας δεν θα επεκταθώ, αλλά έρχεστε εδώ και ε, μας ε, ανεμίζετε φωτογραφίες. Ήταν επίσημη αυτή η παράσταση και δεν ε, εκπροσωπούσα τον εαυτό μου. Είμαι βαθύτατα απογοητευμένος κύριε Έπινγκ. Κύριε Σούλτς, θέλετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να καταθέσω μια προσωπική δήλωση ε, στο τέλος της συζήτησης, όχι μόνο εξ ονόματός μου, αλλά και εξ ονόματος πολλών συναδέλφων που ήταν παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια και παρακολούθησαν τη συζήτηση. Σπάνια, στη διάρκεια της θητείας μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν αισθάνθηκα τόση κακομεταχείριση σε αυτό το παιχνίδι Φαρόμπα ή Μπαρόσο. Εσείς κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας λέτε ε, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που μπορώ να πάρω εγώ. Ότι χάνουν γιατί λέτε τις απορρίπτουν τα κράτη-μέλη και τις αποκρούν. Να σας δώσω τώρα μια συμβουλή να τις καταθέσετε ως νομοθετικές προτάσεις, να δείτε πλειοψηφία θα πάρετε εδώ στο Κοινοβούλιο. Και το Συμβούλιο δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του πλέον. Αλλά και εσείς να μην κρύβεστε πίσω από το Συμβούλιο. Και κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου να σας πω και εσάς το εξής. Έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι στο Συμβούλιο ε, βρίσκουμε συμβιβασμού μεταξύ σοσιαλιστών, συντηρητικών, χριστιανοδημοκρατών και φιλελευθέρων. Κυρίαρχα κράτη συνεδριάζουν στο Συμβούλιο και πρωθυπουργοί. Αποπειράται τώρα ένας πρόεδρος του Συμβουλίου να ανατρέψει και να διαστραβλώσει τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία θεωρίζει ότι το Συμβούλιο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τραβάνε όλο και περισσότερες αρμοδιότητες στον εαυτό τους και μετά επικαλούνται την ομοφωνία. Δεν ήθελε αυτό η Λισαβόνα. Η Λισαβόνα ήθελε λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία και κατά κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρερμηνεύεται κύριε Πρόεδρε τη Συνθήκης Λισαβόνας. Και γι' αυτό έχει φτάσει πλέον η ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει τα ενία στα χέρια του και να ε, υπερασπιστεί μόνο του την κοινοτική μέθοδο. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Πολύ καλά. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς.